So, dear colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Αν δεν έχετε αντίρρηση, εγκρίνεται. Έχω κάποιε σύντομε ανακοινώσει. Η συνεδρίαση θα ακολουθηθεί από τις 6.30 από μια κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών ΕΚΟΝ ΛΥΜΠΕ, όπως γνωρίζετε. Ήδη όμως η αίθουσα έχει και τα καρτελάκια με τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για να μην κάνουμε μετά αναδιευθετήσεις. Οι συστάσει, ε, τα αποτελέσματα των συντονιστών 22 να βρουν στου φακέλου σα και θα σα πω πρώτα ότι σε ό,τι αφορά τα MPL, ε, η διαβούλευση έχετε σύνοψη. Τέλο πάντων, συζητήσαμε και είπαμε ότι η σύνοψη των συζητήσεων και οι δεσμεύσει για την αλλαγή που έγινε στο, ε, στην προσθήκη για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Εξυγίανσης τα βλέπετε σε μια επιστολή που η ΕΚΟΝ λέει ότι θα εφαρμοστούν αυτές οι δεσμεύσεις, μη αυτοματισμός. Δεν θα υπάρχουν γενικά, γενικοί δεσμευτικοί κανόνες, δεν θα υπάρχουν αναβολές, στόκ και θα συνεχίσει ο διάλογος και η συνεργασία στο σημαντικό αυτό θέμα. Επίσης, για το Brexit. Συμφωνήθηκαν το πώς θα προχωρήσουν οι διαπραγματευτές και σε ό,τι την προσωπική επισκέψη στη Βασιλεία θα πάμε τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2018, στη Γαλλία 12 Φεβρουαρίου εκείνη την εβδομάδα του 18 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει ε, μία ε, για την φορολογία και μία για την Τραπεζική Ένωση ε, την εβδομάδα της 18 Φεβρουαρίου και θα δοθούν από τις ομάδες το αργότερο 20 Νοεμβρίου ή τα ονόματα. Το ΕΠΑΡΕΣ θα μας κάνει επίσης μια μελέτη σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις στην συναλλαγματική, συναλλακτική οικονομία, σχέδιο μελέτης για το θέμα του ανταγωνισμού στον τομέα των FinTech, αυτό εγκρίθηκε, σχέδιο προγράμματος εργασιών της ε, ομάδας εργασίας για την Ευσκένα εγκρίθηκε και από εδώ και πέρα τα γραπτά έγγραφα θα δίνονται μόνο στα επίσημα μέλη που ζητούν. Υπάρχει δηλαδή προσέγγιση opt-in για τα έγγραφα, τα γραπτά. Και να το προσέξετε αυτό. Αν δεν το ζητήσετε δεν τα πάρετε γραπτό στα έγγραφα. Πάντως θα υπάρχουν αντίγραφα εφεδρικά, σύμπρεψη κάποιες τα ζητήσει, ό,τι αφορά τον έλεγχο των κατεξότηση υπάρξεων 24 Ιανουαρίου Για το pst 2 θα συζητήσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε πάρει την σχετική κατεξουσιοδότηση πράξη. Κάτι θετικό. Σε ό,τι δεν αφορά την κατεξουσιοδότηση πράξη για την καταπολέμηση του ξεπλήματο χρήματο 22 Οκτωβρίου, η περίοδο συμβουλευτικού ελέγχου παρατείνεται για ένα μήνα, ώστε η Επιτροπή Γιούροβα να μπορεί να έρθει στην ανοιχτή Συνδερίωση των συντονιστών. Και αυτό βέβαια θα λάβει χώρα σήμερα για τη ΜΥΦΙΤ θα σταλεί σε, σε Συμβούλιο και Εκομισιόν ε, επιστολή που λέει ότι ισχύει η τρίμηνη περίοδος κοινοβουλευτικού ελέγχου. Θα υπάρξει και μια ένα ε, σκιωδόν εισηγητών. Σε ό,τι αφορά. Για το ΝΟΝΕ η αναφορά 0296-07 θα στείλουμε στην ε, Επιτροπή των Αναφορών σχετική επιστολή. και για το πρόταση ψηφίσματος δεν θα κάνουμε συνέχεια, δεν θα δώσουμε συνέχεια. Σε ό,τι αφορά το Bank Structure Reform, ε, δεν ε, διαφωνούν οι συντονιστές με την απόσταση πρόταση Κομισιόν. Οι ειδικοί για, το Συμβούλιο δεν είχαμε κάποια αντίρρηση να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε το σχέδιο σύμβασης και για το επόμενο έτος. Συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά ήταν πολλά αυτά που είχα να πω. Περνάμε στο σημείο 3. Όπως ξέρετε, η Κομισιόν έχει προτείνει επαναδιορισμό της κυρίας Ελκε Κένιγκ, θέση του Προέδρου, της Προέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης. Καλώς ήρθατε κυρία Κένιγκ, κυρία Πρόεδρε του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης. Η κυρία Κένικ προεδρεύει από τότε που διορίστηκε το 2014 του ενιαίου Συμβούλου Εξυγίανσης. Η εντολή της ε, έλυγε σύντομα θα λήξει, αλλά θα παραταθεί η θητεία της για την επόμενη πενταετία. Γι' αυτό είναι εδώ σήμερα η κυρία Κένιν. Χαιρόμαστε που είναι εδώ για να μας ε, πει ποια είναι τα σχέδιά της για την επόμενη φάση του Ενίου συμβουλίου έξηγε και πέτυχε στην εναρκτήρια θητεία της. Παρακαλώ, 10 λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ για να σας μιλήσω για τα επιτεύγματα μέχρι τώρα του ενιαίου συμβουλίου υπό την Προεδρία μου και τα στοιχεία που θεωρώ σημαντικά για να προχωρήσει το Συμβούλιο διαφάνεια, η ανάληψη ευθύνη, η λογοδοσία είναι σημαντικά. Στο ρόλο μου ως πρόεδρος είχα συμμετάσχει σε πολλές ανοιχτές και κλειστές ακροάσεις εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και επίσης έκανα και ε, ε, προπαρασκευαστικές επισκέψεις στα συμμετέχοντα κράτη-μέλη και πήγα και σε συνεδριάσεις με εθνικά κοινοβούλια μετά από πρόσκληση γενικά είναι σημαντικό για τους νομοθέτες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλάβουν το ρόλο του Συμβουλίου ε, για την εξυγίαση των τραπεζών και την ε, πρόκληση που αντιμετωπίζει ε, δεδομένου του θετικού αντίκτυπου που μπορεί να έχει η αποστολή του Συμβουλίου στην Ένωση και τους πολίτες. Εμείς δημοσιεύσαμε το πρώτο πρόγραμμα πολιετές για τα επόμενα τρία χρόνια και το πρόγραμμα μας για το 2018 σήμερα και ήδη μπορούμε να πούμε ειλικρινώς ότι ο δεύτερος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης εδράζεται σε στέρεα θεμέλια, αλλά πρέπει την δυναμική να τη συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε και να παράσχουμε και να υλοποιήσουμε τους φιλόδοξους στόχους που έχουν τεθεί από τους συνομοθέτες, ε, που δεν είδε να έχει ολοκληρωθεί η αποστολή μας ακόμα. Τα επόμενα χρόνια το Συμβούλιο Εξυγένσης θα συνεχίσει να θέτει τις προϋποθέσεις και να προχωρεί σε τακτική εξυγίανση των τραπεζών που έχουν προβλήματα με ελάχιστο αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία και τα δημόσια οικονομικά. Αυτή είναι η αποστολή μας και ε, αυτό είναι ένα πρόγραμμα, ένα έργο πολυετές, επειδή έχει πολλές πτυχές και συνθετότητες. Συγκεκριμένα, στο τέλος του, μέχρι το 2020 το αργότερο, σίγουρα για τις μεγάλες τράπεζες πιο νωρίς, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα έχει αναπτύξει πλήρη προγράμματα εξυγίανσης για όλους τους τραπεζικούς ομίλους, προγράμματα με μεγάλη εκλέπτυνση στο πλαίσιό μας. Εμείς θα έχουμε και ενδιάμεσα στάδια για τα σχέδια εξυγίανσης τα οποία θα βελτιωθούν σταδιακά μέχρι να φτάσουν το τελικό στάδιο. Διευκρινίζω ότι ήδη έχουμε σχέδια για την συντριπτική πλειοψηφία των τραπεζών μας. Τώρα πρέπει να τα βελτιώσουμε, να τα εμπλουτίσουμε. Και επίσης, όπως και σε άλλους τομείς της ζωής, πρέπει να πω ότι το σχέδιο είναι καλό στο βαθμό που μπορεί να αντιμετωπίσει μια άγνωστη πραγματικότητα τα προγράμματα, τα σχέδια ε, προσανατολίζονται προς το μέλλον, αλλά αναπόφευκτα θα πρέπει να προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες συνθήκες, όποτε και αν θα ε, περάσουν σε σχέδιο εξυγίανσης και συνεχώς πρέπει να αναβαθμίζονται, να ανανεώνονται και να ενημερώνονται, δεν μπορούν να μένουν στάσιμα. Ε, το... Μέχρι τότε λοιπόν θα έχουμε ε, ε, στόχους δεσμευτικούς με ελάχιστες προϋποθέσεις για τα, ε, τα, τα, ίδια κεφάλαια και τις υποχρεώσεις της επιλέξιμες και αυτό θα βοηθήσει να φύγουν τα εμπόδια στην εξυγίανση. Για τους τραπεζικούς ομίλους με έναν συνάδελφο τα σχέδια για το 2017 συμπεριλάβουν δεσμευτικούς στόχους ε, σε ενοποιημένο επίπεδο, όπως και μια αρχική συζήτηση των, των στόχων αυτών ε, σε επίπεδο ουσιαστικό. Ε, αν δεν υπάρχει σχέδιο εξυγίανσης, θα ορίσουμε σχέδια επιλέξιμο, ιδίων πόρων και επιλέξιμων παθητικών. Έχουμε ήδη παρουσιάσει την, ε, τα σχέδιά μας σε δύο διαλόγους του κλάδου το 2017. Το 2018 για τις τράπεζες όπου υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι φέτος σε ενοποιημένο επίπεδο το ε, Συμβούλιο θα καθορίσει σε εξατομικευμένο, ε, εξατομικευμένο επίπεδο του στόχου. Συνεχίζομαι. Για τους άλλους θα θέσουμε στόχους σε ενοποιημένο επίπεδο δεσμευτικούς. Η προσέγγιση διασφαλίζει ότι οι τράπεζες θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη μεταβατική περίοδο για να αντιμετωπίσουν τις προϋποθέσεις χωρίς μεγάλο αντίκτυπο στη δημοσιονομική, χρηματοπιστωτική ε, σταθερότητα, την οικονομία ή την δανειοδοτική τους ικανότητα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν αποφασίστηκε το πλαίσιο εξυγίανσης υπήρχε συνένεση ούτω ώστε να μην αποφύγουμε αυτά που έγιναν κατά την χρηματοπιστωτική κρίση. Να χρησιμοποιήσουμε χρήματα των φορολογουμένων για να διασώσουμε τις τράπεζες επειδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Ε, ε τώρα πιστεύω ότι, θα, ε, ότι έχουμε σχεδιάσει ένα εργαλείο το οποίο θα αντιμετωπίσει αυτούς τους κινδύνους, ε, θα αντιμετωπίσει δηλαδή με διαφορετικό τρόπο τα πράγματα, όχι σε βάρος των ε, φορολογουμένων. Ε, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι είναι, πολύ, είναι στην καρδιά των στόχων μας ε, όλα αυτά, όπως ήταν και στην χρηματοοικονομική κρίση του 2008, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι τράπεζες στην Τραπεζική Ένωση ε, εξέδωσαν πολύ περισσότερα additional tier 1, 2 και ε, unsecured bonds, senior unsecured bond, το πρώτο μισό του 2017 από ότι το δεύτερο μισό του 2016. Οπότε πάμε καλά αν και δεν υπάρχουν παντού δεσμευτικοί στόχοι. Το Συμβούλιο θα προχωρήσει τις κοινέ πολιτικές εξυγίανσης και τα πρότυπα σε τομείς κλειδιά το 2018. Για παράδειγμα, θα αναπτύξουμε πολιτικές σχετικά με τα εσωτερικά MRL, τη διαβάθμιση των MRL για ε, στρατηγικές ε, ε, και ε, ρευστότητας κατά την εξυγίανση. Ε, επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σοβαρά εμπόδια και του χρόνου θα επικεντρωθούμε στον εντοπισμό των εμποδιών αυτών και θα αντιμετωπίσουμε ότι και θα αναθέσω μέσα στις τράπεζες να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης ε, θα πρέπει να δούμε τα διάφορα εργαλεία για την εξυγίανση και την αξιολόγηση του δημοσίου συμφέροντος που είναι καυτό θέμα κατά την εξυγίανση. Ε, περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο έγγραφό μας για τον πολιετή προγραμματισμό μας όπου τα παρουσιάζουμε όλα αυτά. Η ανάληψη δράση εξυγίανση χρειάζεται ένα γενικό σχέδιο για τα διαφορετικά σενάρια. Είχαμε τον Ιούνιο την πρώτη περίπτωση, την πρώτη α, ε, υπόθεση μετά την αξιολόγηση της ε, ΕΚΤ ότι η Banco Popular ε, είχε πρόβλημα και το Συμβούλιο μαζί με την Εθνική Αρχή Εξυγένσης της Ισπανίας προχώρησε να, σε εξυγένση της Banco Popular. Το ε, Συμβούλιο μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ θα λάβει υπόψη τα διδάγματα που αντλήσαμε από αυτή την εμπειρία της εξυγίανσης. Όμως, ε, όποιο μοντέλο κρίσης παρουσιάσουν οι καλύτεροι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να ε, αξιολογήσουμε την πραγματικότητα που μπορεί να είναι διαφορετική σε κάθε περίπτωση και θα πρέπει να δράσουμε με δεξιοτεχνία και ευελιξία όταν πρόκειται για προβληματικές τράπεζες και την εξυγίανσή τους, δεν υπάρχει ε, δυστυχώς δεύτερη ευκαιρία. Μπορούμε να πάρουμε την περίπτωση της Banco Popular ως παράδειγμα, ε, όπου είχαμε, ε, είχαμε προβλέψει και τον Μπέιλιν ως ενδεχόμενο, αλλά μπορούμε να πούμε ότι τώρα λαμβάνοντας υπόψη ότι επειδή είχαμε δυνητικό αγοραστή για όλη την τράπεζα, είχαμε αυτή την τύχη Οπότε μπόρεσαν οι λειτουργίες να συνεχιστούν και αν, όπως ε, γίνεται εδώ, ε, ε, αν υπάρξει αυτή η εναλλακτική, αυτή είναι η προτιμόμενη, όπως σε αυτή την περίπτωση, ανεξάρτητα από τα άλλα. Οι παρεκκλήσεις θα πρέπει βέβαια να εξετάζονται αν δώσουν καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, αναπόφευκτα η εξυγίανση οδηγεί σε ζημίες για τους κατόχους για τους μετόχους και τους κατόχους τους ομολογιούχους. Εμείς ε, θα πρέπει, ε, να, έτσι όπως το βλέπουμε, να λάβουμε υπόψη μας και τη δράση των δικηγόρων που προσβάλλουν όχι μόνο τις δράση της Ένωσης και των εθνικών αρχών, αλλά και την ομιμότητα του πλαισίου εξυγένσης της Ένωσης. Ε, θα, τα επόμενα χρόνια θα δούμε αλλαγές, αλλαγές που θα πρέπει να τις αποφασίσετε. Και πράγματι η εξηγένση των τραπεζών είναι καινοφανέ εργαλείο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με βάση τους υφιστάμενου κανόνε, λαμβάνοντα υπόψη εσωτερική εμπειρία που έχει ε, αντληθεί και στο βαθμό που δεν ε, ε, ε, οδηγεί σε λανθασμένες αποφάσεις. Θα πρέπει να, δούμε και το, την άλλη πλευρά του πακέτου που είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζομαι ότι θα ε, εντείνει το πλαίσιο της εξυγίανσης και θα διευκρινίσει την πολιτική μας τα επόμενα χρόνια. Πριν ολοκληρώσω θα ήθελα να πω ότι η εφαρμογή του κοινού backstop για το, το ε, ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης ε, είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να στηρίξουμε τις προσπάθειες των κρατών μελών για να δημιουργήσουν αποτελεσματικό κοινό backstop. Τέλος, πάντα το λέω αυτό στο τέλος, ε, το έντις είναι ο τρίτο πυλώνα τη Τραπεζική Ένωση και ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί. Ε, γενικότερα θα υπενθύμιζα στα κράτη-μέλη την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε θέματα ε, legacy ε, του, του, του, του, ιστορικού παρελθόντος και να βελτιώσουν το νομικό πλαίσιο. Ε, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να εδραιώσουμε το έργο που έχει γίνει τώρα στο σχεδιασμό των εξηγιάνσεων και να εμβαθύνουμε την ανάλυση μας και ίσως ό,τι αφορά το σχεδιασμό της εξυγένσης και την πολιτική ανάπτυξη. για να συνοψίσω, πολλή εργασία έχει γίνει ήδη, αλλά ακόμα δυστυχώ, δεν μπορούμε να δηλώσουμε ότι η αποστολή μας έχει ολοκληρωθεί. Ελπίζω να γίνει αυτό. Ε, ε, ελπίζω να συνεχίσω με το έργο αυτό στο μέλλον και ευχαριστώ για την προσοχή σας και την υπομονή σας. Προσπάθησα να τηρήσω το δεκάλεπτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα αρχίσουμε με τις ερωτήσεις ή σχόλια. Ο Μπράιν Χέις από το ΕΛ. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και η κυρία Κένιγκ. Σας καλωσορίζουμε στην ΕΚΟΝ και ευχαριστούμε για την εισήγησή σας. Στο τέλος αναφέρατε τι πρέπει να κάνουμε, διότι πρόκειται για μια εργασία εν εξελίξη. Μιλήσατε για το ίντις που είναι το, ο τρίτος πυλώνας της ε, Τραπεζικής Ένωσης και μιλήσατε και για την ανάγκη να βελτιώσουμε τα επίπεδα αφαιρεγγιότητας στα κράτη-μέλη. Πρέπει να γίνουν πολλά, λοιπόν. Σε περιβάλλον λειτουργίας του Συμβουλίου Εξυγίανσης θα πρέπει να δούμε ότι έχουμε το σωστό μείγμα πολιτικό. Και μετά την κρίση δεν ξέρω κατά πόσο η εξυγίανση αυτή των τραπεζών κινείται προς τη διάσωση με ίδια μέσα και όχι διάσωση με δημόσιους πόρους. Αυτό είναι ύψης της σημασίας και αυτό που κάνατε τα προηγούμενα χρόνια θα οδηγήσει σε μια μελλοντική εργασία έτσι ώστε να υπάρχει η εμπιστοσύνη του κοινού προς μια πραγματική εξυγίανση με βάση και τη λειτουργία της ΕΚΤ. Θεωρείτε ότι μπορεί να βελτιωθεί η σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν ναι, πώς έρχεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα ενώπιών μας αλλά μέσα στα πλαίσια της συνιστώσας της διαφάνειας για την ε, λειτουργία του Συμβουλίου Εξυγίανσης, τι μπορεί να γίνει και επίσης δεν είδα το πολιετές σχέδιο που δημοσιεύτηκε σήμερα, το οποίο καλωσορίζω. Πώς θεωρείτε όμως ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα μέρη του κόσμου όταν μιλάμε για ε, ε, σχέσεις ε, ρευστότητας και προαπαιτήσεις για εξυγίανση. Τι μπορούμε να κάνουμε το πακέτο αυτό εργαλείων αρκεί και ε, θα ήθελα και χαίρομαι μάλλον που θα συνεργαστείτε με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα τα υποδεχτείτε μέχρι το τέλος της θητείας. Νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα που μπορείτε να αποστείλετε στα μεγάλα και τα μικρά κράτη-μέλη, έτσι ώστε να ενθαρρύνεται αυτό τον διάλογο, κάτι το οποίο καλωσορίζω. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Αρχίζοντας από την τελευταία ερώτηση. Χαίρομαι για την ανταλλαγή απόψεων με όλα τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά θα μεταβώ όταν προσκληθώ φυσικά. Θέλουμε φυσικά να προωθήσουμε αυτό το διάλογο το Συμβούλιο Εξυγίανσης δεν πέτυχε τα τρία πρώτα χρόνια να επισκεφθεί κάθε κράτος μέλος για να μιλήσει με τη βιομηχανία, με τα, το θησαυροφυλάκιο και ούτω καθεξής. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας, Έχουμε όμως ορίσει συναντήσεις με συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Εν πάση περιπτώσει θα προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων και με τα Εθνικά Κοινοβούλια, εκεί που απαιτείται. Υπάρχει πολύ καλός διάλογος με τις ΗΠΑ και με την Τράπεζα της Αγγλίας, ένα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι της Τραπεζικής Ένωσης και επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει αν αποτύχουμε σε, εν, σε μία από τις συνιστώσεις μας. Και οι, τα άλλα μέρη έχουν να αντιμετωπίσουν ένα κράτος, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη είπα και ούτω καθεξής. Εμείς έχουμε 19 διαφορετικούς νόμους περί αφαιρεγγιότητας και εταιρικούς νόμους. Άρα η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη. Όλοι όμως αντιμετωπίζουμε τα ίδια ζητήματα. Πρόκειται για δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι πολύ πιο δύσκολο όταν μιλάμε για την εξυγίανση σε, επίπτωση, σε περίπτωση ρευστότητας, διότι εδώ μιλάμε για την Bank of England, για την Fed, και στη δική μας περίπτωση με την ΕΚ. Θεωρώ ότι οι σχέσεις μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ καλές. Προσπαθούμε να υπάρχει διαφάνεια, να έχετε πρόσβαση στα πρακτικά μας και πάντα ήμουν ανοιχτή για συναντήσεις. και αυτό σε επίπεδο της δικής σας επιτροπής ή και κλεισμένων των θυρών. Πρόκειται για κάτι το οποίο ε, παίρνω υπόψη και εκτελώ πολύ σοβαρά. Περβάνς Μπερές. Ευχαριστώ την ε, Έλκε Γκάνιγκ. Η και κλεισμενων των θυρων προκειται για κατι το οποιο παιρνω υποψη και εκτελω πολυ σοβαρα περβανος μπερες ευχαριστω την ελκε γκανιγκ η ανανεωση της θητείας σας στο ενίο Συμβούλιο Εξυγίανσης λαμβάνει χώρα τη στιγμή που πολλοί φορείς της αγοράς κοιτούν εκ του σύνεγγυ στην κατάσταση γιατί χρησιμοποιήσατε την εργαλειοθήκη της εξυγίανσης. Εμείς θέλουμε να υποβάλουμε πληθώρα ερωτήσεων προς όλες τις κατευθύνσεις. Μέσα στα πλαίσια αυτής της κοινοβουλευτικής νομιμότητας, λοιπόν, μπορούμε να αποτιμήσουμε την κατάσταση με τη ε, εξυγίανση της Banco Popular ή των Ιταλικών τραπεζών. Ως πρόεδρος του Εννέου Συμβουλίου Εξυγίανσης θα ήθελα να σας ρωτήσω πέρα από αυτά που είπατε με τη διαχείριση ρευστότητας θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι, ποια είναι τα σφάλματα που έγιναν στο παρελθόν, ιδιαίτερα τις πληροφορίες που δόθηκαν στις αγορές πριν από το Συμβούλιο, πριν να αποφαθεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση ας πούμε της Banco Popular. Μιλήσατε επίσης επί μακρόν για πληθώρα θεμάτων και θα ήθελα να ρωτήσω πώς ε, οι τράπεζες μπορούν να πάνε στις αγορές για να αποκτήσουν νέα στοιχεία ενεργητικού χωρίς να υπάρχει μία κυκλική πορεία η οποία καθιστά την αγορά κεφαλαίου πιο ακριβή. Μιλήσατε για τετράχρονη στρατηγική, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω πώς θα επιλύσετε αυτή την αντίφαση, δηλαδή να λάβετε υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε τράπεζας χωρίς να αυθαιρετείτε. Ως προς την ΕΝΤΙΦ, όλοι μας ε, γνωρίσαμε, ε, γνωρίσαμε την κατάσταση μετά την ε, πτώχευση της Banco Popular και ευτυχώς βρέθηκε αγοραστής. Θεωρείτε ότι η τακτική επικοινωνίας και ανακοινώσεων της Επιτροπής οδήγησε σε εξέλιξη της κατάστασης ή όχι. Όμως η μείωση των κινδύνων ισχύει αλλά μέχρι πόσο, μέχρι πού πρέπει να μειώσουμε τους κινδύνους, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στον επιμερισμό ε, ευθυνών και κινδύνων, ανάληψης ε, κινδύνων. Θα προσπαθήσω να απαντήσω τις ερωτήσεις σας. Στην ε, περίπτωση της Banco Popular είπαμε ότι είχαμε να κάνουμε με μία περίπτωση όπου θα έπρεπε να ισχύσουν οι κανόνες κατά γράμμα, αλλά ευτυχώς υπήρξε αγοραστής και ήμασταν πολύ τυχεροί διότι η ίδια η τράπεζα είχε προταθεί προς πώληση, είχε αυτοπροταθεί προς πώληση και αυτό στοιχειοθέτησε την εργασία μας. Γι' αυτό είπαμε στη συνέχεια ότι δεν πρόκειται για σφάλμα, αλλά και αυτή η περίπτωση έδειξε ότι το θέμα της ρευστότητα και της εξυγίανσης έχει μεγάλη σημασία και εδώ είχαμε δεδομένα τα οποία οποία ε, εξετάσαμε και η τράπεζα μας έδωσε τις πληροφορίες που θέλαμε, αλλά έπρεπε να δώσει μεγάλο αγώνα εάν χρειαζόταν ε, μεγαλύτερη διαφάνεια για το κύριο χρέος. Γι' αυτό τα δεδομένα είναι ύψης της σημασίας. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει μία διαδικασία πώληση της τράπεζας, υποπίεση χρόνου είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί αγοραστής ε, για την τράπεζα. Το δεύτερο, μιλήσατε για τις πληροφορίες προς τις αγορές δεν υπήρξε διαρροή πληροφοριών από εμάς προς την αγορά, προς τις αγορές. Ήταν γνωστό ότι η τράπεζα είχε υποστεί πιέσεις και ε, το Reuters είναι αυτό που θα ε, πει ποιος ε, έδωσε τις πληροφορίες. Το ΜΡΕΛ, δηλαδή οι ελάχιστες απαιτήσει ιδίων κεφαλαίων και αποδεκτών υποχρεώσεων, το ΜΡΕΛ λοιπόν θα πρέπει να αφορά ε, συγκεκριμένα ποσά, τάξεις μεγέθους δηλαδή, και γίνεται μία συζήτηση επί του παρόντος. Αποφασίσαμε και αυτό έχει δημοσιοποιηθεί στον ιστό τοπό μας, ότι υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι μέχρι τέσσερα χρόνια για συμμόρφωση. Μερικές ε, τράπεζες έχουν ήδη συμμορφωθεί, άλλες όμως χρειάζονται την τετραετία. Αλλά το ΜΡΕΛ, δηλαδή οι ελάχιστες απαιτήσει ιδίων κεφαλαίων, θα πρέπει να μας απασχολήσει σε ετήσια βάση. Η, ως προς την έντις είπαμε ότι υπάρχουν τρία επίπεδα και το τρίτο επίπεδο είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε να υπάρξει τραπεζική ένωση, πραγματική τραπεζική ένωση έτσι ώστε το θέμα να μην φτάσει στους καταθέτες που αποτελεί εθνικό εγχείρημα. Θεωρούμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε στην σωστή κατεύθυνση για το τι μπορούμε να συζητήσουμε εδώ, Σάντερ Λούις. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Κένιγκ. Έχω κάποιες ερωτήσεις ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και το έντις. Ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις είναι και η στιγμή ε, να μας πείτε αν έχετε ένα δώρο που θα θέλατε να λάβετε ε, τα Χριστούγεννα. Να αλλάξουν κάποιοι κανόνες ή όλα λειτουργούν καλά. Η εικόνα είναι ροζ ή όχι. Ρόδινη. Θα πρέπει μήπως να αναθεωρηθεί η πρόταση για τις κρατικές ενισχύσεις του τραπεζικού τομέα, το BRRD, να ευθυγραμμιστεί. Και το δεύτερο για το έντι στο σύστημα καταθέσεων Δύο χρόνια συζητάμε ένα πλήρω ανεπτυγμένο σύστημα, το είπατε και στην εισαγωγή σας και απαντώντα σε συνάδελφο Πέρβανς Μπερέ, έχω ένα ερώτημα για το ρόλο των εθνητών αποθετικών ε, συστημάτων ε, εγγύης καταθέσεων. Μιλάτε για μικρές ε, τραπεζικές συναλλαγές που μπορεί να μην χρειάζεται να υπάρχουν ευρωπαϊκά ταμεία που θα παρεμβαίνουν, είναι, ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση στο πλαίσιο του έντηση τι πρέπει να γίνει και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν θεωρείται ότι πρέπει να υπάρχουν αυτά τα εθνικά συστήματα και να μπορεί να υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης ε, των απολειών και στο τελικό στάδιο ε, είναι κάτι το οποίο μπορείτε να το υποθέσω ότι θα γίνει πραγματικότητα ναι, για το ευχολόγιό μου που πράγματι επειδή τα Χριστούγεννα είναι επίκαιρο θα μπορούσα να πω ότι μετά την εξυγίανση ε, αφαιρι... περιπτώσεων που είδαμε κατά το παρελθόν. Λογικό θα ήταν, πιστεύω, με τι απαιτούμενε εγγύσει και για βέβαια, να δούμε μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε μία δέσμη κινήτρων θα τα χαρακτηρίζα εγώ. Δηλαδή, να έχουμε ε, το banking communication, αναφερήθηκε το 2013 τελευταία φορά, Έχουμε τον BRD 2014, οπότε λογικό θα ήταν ε, να αναθεωρηθούν για να ευθυγραμμιστούν αυτά τα δύο το ένα με το άλλο. Να είμαι σαφής τώρα. Εγώ δεν είμαι αυτή που θα πω ότι δεν χρειάζεται η ε, προφυλακτική ανακεφαλοποίηση. Θα πρέπει να το έχουμε αυτό ως ε, εργαλείο στην αρελευθερική μας και η παροχή βοήθειας για την εξήγηση. Και αυτό θα μπορούσε να είναι λογικό. Απλά θα πρέπει να υπάρξει ευθυγράμμιση. Δηλαδή, να μην ε, μπορεί κανείς ε, να ευνοηθεί με το ένα ή το άλλο σενάριο περισσότερο για εθνικά συστήματα αγγίσκα φυσικά και θα πρέπει να έχουν ρόλο στο μέλλον στο πλαίσιο του ε, της εμείς είμαστε το Συμβούλιο Εξηγίασης, ε, αρμόδιοι για τις μεγαλύτερες τράπεζες αλλά συνεργαζόμαστε στενά με τις εθνικές αρχές εξηγίανσης, που είναι οι αρχές εξηγίανσης, για τις μικρότερες τράπεζες που έχουμε εκεί μόνο μία ελεγκτική δράση, το έντις επίσης πάντοτε, θα είναι ένα θέμα που θα εστιάζει κυρίως στα εχέγγυα για τις μικρομεσαίες τράπεζες δεν είναι ευρωπαϊκές, ε, ως προς την εποπτεία δηλαδή, δεν εποπτεύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή υπάρχουν εθνικές αρμοδιότητες και ευρωπαϊκές αρμοδιότητες στο σύστημα εξυγίανσης αλλά αυτό το βλέπω ίσως για πιο μετά. Είναι λίγο νωρίς να το συζητήσουμε από τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε κυρία Κέννη και συγχαρητήρια για την ε, ανανέωση της θητείας σας. Και εγώ θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία σημερινή ακρόαση για να δούμε τι γίνεται με την ανάκαμψη και το πλαίσιο εξυγίανση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς έχουν αποδώσει. Θα ήθελα να εστιάσω στην έννοια του δημόσιου συμφέροντος, public interest, που είναι στο επίκεντρο. Και επανέρχομαι σε δύο πρόσφατες υποθέσεις ταλικών τραπεζών που έπρεπε το δημόσιο να επομιστεί μέρος των βαρών. Εφαρμόστηκαν εθνικοί κανόνες αφαιρεγγιότητας και όχι οι ευρωπαϊκοί κανόνες bail-in. Και έχω το εξής ερώτημα, τα εξής ερωτήματα. Πρώτον, αν η εφαρμογή των εθνικών κανόνων αφαιρεγγιότητας δημιουργεί έξοδα για το φορολογούμενο, όπως έγινε με τις δύο τράπεζες της Ιταλικές από τη Βενετία. Δεν θα ήταν καλύτερο να εφαρμοστεί αντίθετα το BRRT. Και δεύτερον, αν το δημόσιο συμφέρον ορίζεται ως η διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ε, η Ιταλική κυβέρνηση πώς και ζήτησε και είπε πολύ καιρό ότι ε, έπρεπε να θεωρηθούν συστημικές αυτές οι Ιταλικές τράπεζες. Αλλά τελικά ε, διαφορετικό ήταν το συμπέρασμα. Είναι λίγο απόρρια άξιον αυτό, γιατί το έχει πει ξεκάθαρα η κυβέρνηση ότι χρειάζονται μέτρα αφαιρεγκαιότητα για να αποφευχθούν σημαντικέ ταράξει στην οικονομία. Τέλο, συμφωνείτε ότι το δημοσιοφέρον θα μπορούσε να οριστεί κατά κάποιο τρόπο και ω ε, το μέτρο αξιοπιστία των κανόνων. Για τι δύο αυτέ τράπεζε, παραλαμβάνω, Μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι οι κανόνες ερμηνεύτηκαν με κάποια διακριτική ευχέρεια. Ευχαριστώ. Απάντηση. Για το πλαίσιο BRRD, οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση. Εκεί προβλέπεται ότι αν έχουμε μια προβληματική τράπεζα που καταραίει, πρώτον πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει η ιδιωτική λύση ήταν αναπόφευκτο στην προκειμένη περίπτωση, ε, το προσπάσαν δεν υπήρχε δυτική λύση. Δεύτερον, ελέγχουμε αν υπάρχει δημόσιο συμφέρον για την εξυγίανση των τραπεζών στο πλαίσιο του BRRD, της οδηγία αυτή, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμοστεί το εθνικό πλαίσιο αφαιρεγκαιότητα. Δημόσιο συμφέρον λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Από τα πέντε κριτήρια Δύο λαμβάνουμε ιδιαίτερα υπόψη μας. Το πρώτο είναι κατά πόσον υπάρχει απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και το δεύτερο κριτήριο είναι εάν τράπεζες ή η τράπεζα παρέχει κάποιες κρίσιμες λειτουργίες. Αυτά είναι τα βασικά που πρέπει να ελέγξουμε. και άλλα, αλλά αυτά είναι τα βασικά. Για τις δύο τράπεζες που αναφέρατε, θεωρήσαμε ότι λόγω της μεγάλης απομόκληση που είχε γίνει στις δύο αυτές τράπεζες, σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε κάποια κρίσιμη λειτουργία που δεν θα μπορούσε να υποκατασταθεί. Ούτε επίσης διαπιστώθηκε ότι ήταν διασυνδεδεμένες με τη βιομηχανία και θα μπορούσε αυτό να οδηγήσει σε χρηματοψηφιστική αστάθεια. Άρα θεωρήθηκε ότι στην προκειμένη περίπτωση οι εθνικέ αρχέ πρέπει να αναλάβουν την ε, ε λύση του προβλήματο. και εφαρμόστηκαν εθνικοί κανόνε αφαιρεγκαιότητα και η σχετική νομοθεσία. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Εκεί μιλάμε για απόλυση της επιχείρησης. Αυτό ήταν το ε, αποτέλεσμα. Η απόφαση της Ιταλικής κυβέρνησης ελήφθη σε διαβούλευση και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήταν να δοθεί βοήθεια όχι λόγω δημοσιοσυμφέροντος για τη σταθερότητα συνολικά στην Ιταλία αλλά το επίκεντρο ήταν κοινωνικές κυρίως πτυχές και πολλές άλλες πτυχές στην Ιταλία. Εμείς είχαμε λάβει πριν μια απόφαση, δεν είχαμε περιθώρια, αλλά αυτό έρχεται στο έρθμα του κύριου Λούντς λίγο για το ευχολογιό μας και τι θέλουμε και εμείς θέλουμε να σκεφτούμε και τις υποθέσεις αυτές μαζί με την Κομισιόν να μελετήσουμε τις υποθέσεις για να δούμε χρειάζεται ευθυγράμμιση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βιέγκας. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Έχω ορισμένες ερωτήσεις σε σχέση με το παρελθόν και τα παρελκόμενά του. Σε σχέση με το Banco Popular της Ισπανίας, θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουν εκφραστεί, έχουν υποβληθεί πολλές προσφυγές ενώπιον της δικαιοσύνης, κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια γενική παραλυσία. Δεύτερον, σε σχέση με την διαρροή πληροφοριών, που έδωσε το Reuters στις 31 Μαΐου, θα ήθελα να πω ποια ε, είναι τα διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε. Πόσο οδήγησε αυτή η διαρροή σε μία κρίση, ε, κρίση ρευστότητας της τράπεζας. Ως προς την τράπεζα αυτή, η Deloitte έπρεπε να υποβάλει δύο ε, εκθέσεις, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων, που δείχνει ότι υπάρχουν πολλές ασαφίες και ευαλωτότητες σε σχέση με σύγκρουση συμφερόντων. Αυτά ορίζει η πρώτη έκθεση της Deloitte. Και δεύτερον, ως προς την ε, διαφάνεια, Πότε θα μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στις δύο αυτές εκθέσεις και κατά πόσο μπορούμε να μιλήσουμε για το ίδιο κριτήριο διαφάνειας. Δηλαδή, ε, διατρέχουμε τον κίνδυνο να έχουμε μία κατακαιρματισμένη έκθεση τη στιγμή που και στις δύο εκθέσεις υπάρχουν στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα. Άρα, αυτή η εξωτερική ανάθεση ε, δεν καθιστά πιο ευάλωτο το σύστημα. Είναι επίγον το σύστημα εποπτείας να διαθέτει ε, μέσα ανεξαρτησίας και ανεξάρτητης κρίσης αυτών των επιχειρήσεων τύπου Deloitte που αποτελούν ή μάλλον λειτουργούν εν είδη ολιγοπολίων. Η εξυγίανση οδηγεί σε συγκέντρωση, σε συγκεντρωτισμό του χρηματοπιστωτικού συστήματος και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό αποτελεί η προτεραιότητα της Ταπεζικής Ένωσης καθεαυτής πολλές ερωτήσεις. Θα τις απαντήσω μία προς μία. Οι καταγγελίες ε, δεν θα σταματήσουν την εξυγίανση, δεν μπορεί δηλαδή να ανασταλεί η απόφαση. Η νομοθεσία προβλέπει ότι αν, και ελπίζω να μην συμβεί αυτό, είμαι πεπισμένη μάλλον δεν θα συμβεί, όταν και ε, αν η εξυγίανση ε, παραβιάζει νομοθεσία, αν κάποιος ε, ομολογιούχος διατρέχει κίνδυνο, ε, τότε θα υπάρξει αποζημίωση και το ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης θα δώσει την αποζημίωση αυτή. Αυτά σε γενικές γραμμές. Όχι λοιπόν, δεν μπορεί να ανασταλεί η απόφαση εξυγίανσης. τώρα, ποια μέτρα θα ληφθούν ε, νομίζω ότι πάντοτε έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να υπάρχει ενημέρωση σε όλους, σε κάποιον οργανισμό και σίγουρα είναι απόλυτη ανάγκη να φροντίσουμε ότι τα δεδομένα θα είναι εμπιστευτικά μέσα στον οργανισμό. Να επαναλάβω όμως ότι αυτή είναι μία έκθεση που υποτίθεται ότι βγήκε από μας ενώ δεν έχει βγει από μας. Τώρα, ε, ε ε, ποιο, αν αυτό ήταν το σημείο που ήταν καταλήτης, όχι υπήρχαν προβλήματα, ε, υπήρχαν ε, αξιολογήσεις αρνητικές. Θα ήταν πολύ εύκολο να πούμε ότι οι Reuters έδρασαν καταλήτικα. Η έκθεση Deloitte, εξάντε εξ των προτέρων εκ των υστέρων, εδώ Ποιος ε, θα πρέπει να κάνει την αξιολόγηση. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη. Θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση από ανεξάρτητο τρίτο μέρος. Γι' αυτό το Συμβούλιο Εξυγίανσης ήδη το 2015 ε, έκανε ε, ενέργειες ούτως ώστε να έχουμε τους συνήθεις υπόπτους, έξι εταιρείες συνολικά που συμμετείχαν και διασφαλίσαμε ότι όταν ετοιμάζουμε εξυγίανση και στην περίπτωση της Banco Popular εμείς θα πρέπει να δούμε τη σύγκρουση των συμφερόντων, θα το ελέγξουμε το θέμα αυτό και μετά θα επιλέξουμε μια εταιρεία που θα ε, μας δίνει την καλύτερη προσφορά για τη δουλειά που θέλουμε. Και υπάρχουν, υπήρχαν δύο διαφορετικές, ε, γίνονται δύο αξιολογήσεις. Μία θα ενημερώσει εμάς σχετικά με το πλαίσιο και τα εργαλεία εξυγίανσης που θα δώσουν υποθέτω με τα καλύτερα αποτελέσματα και μετά εξπόστε γίνεται η αξιολόγηση ε, πάλι των στοιχείων για να βεβαιωθούμε ότι κανένας πιστωτής δεν θα είναι σε χειρότερη θέση ε, από ότι αν δεν είχε, δεν είχε γίνει η εξυγίανση. Τώρα, είναι καλύτερα να γίνει εσωτερικά και να έχουμε ένα στρατό προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη ότι είμαστε 19 κράτη-μέλη και θα πρέπει να, είμαστε, να έχουμε την καλύτερη ενημέρωση για να γίνει σωστή αξιολόγηση. Το νομικό πλαίσιο δεν το έχει απαντήσει αυτό. Λέει ότι θέλουμε να είναι ανεξάρτητη τρίτη εταιρεία. Για τη διαφάνεια, μετά την εξυγίανση δημοσιεύσαμε ε, την ε, απόφαση ε, εξυγένσης. Το Συμβούλιο της, του, το Διοικητικό μας Συμβούλιο θεωρεί ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την έκθεση αξιολόγησης. Η έκθεση αξιολόγησης θα πάρει κάποιες βδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα για την δεύτερη αξιολόγηση. Γιατί η τρίτη αξιολόγηση ακόμη δεν έχει δημοσιευτεί, δεν έχει φύγει από τα χέρια του αξιολογητή και δεν τους πιέσαμε γιατί θέλουμε να είναι πλήρης, θέλουμε να είναι ακριβείς και να μην μπορούν να μας πούν ότι μας πιέσατε πολύ και δεν είμαστε τέλειοι. Ε, όταν τη λάβουμε θα κάνουμε την ίδια διαδικασία και για την τρίτη αξιολόγηση. Και για τη συγκέντρωση του συστήματος, οι συγχωνεύσεις οδηγούν σε συγκεντρώσεις. Αλλά το too big to fail ε, είναι κάτι παραπάνω από ένα στοιχείο μεγέθους. Ευχαριστώ, Σβεν Γκίγκολτ. Ευχαριστώ. Καταρχήν για την Banco Popular Ήδη έχουμε ενδελεχώς συζητήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν και εκφράσαμε τις ανησυχίες μας. Σίγουρα είναι θεμητό δικαίωμα οποιοδήποτε χάνει χρήματα σε αυτή την περίπτωση να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλο λόμπινγκ και εδώ στο Κοινοβούλιο και αλλού. Και αυτό θεωρώ ότι συνιστά πρόβλημα πως κάποιοι καλά οργανωμένοι δρόντες βάζουν το θέμα ε, στην ημερήσια διάταξη και επιτάπητος. Πείτε μας περισσότερες λεπτομέρειες. Τι πιέσεις είδατε εσείς να υπάρχουν ε, και σας απειλούν. Τι αντιμετωπίσατε. Δεύτερον, σχετικά με την επικείμενη ψηφοφορία. Θα ήθελα γενικά να πω ότι έχουμε την αίσθηση ότι στα κράτη-μέλη, στην κοινή νόμοι και εδώ ε, υπάρχει διάθεση για σκληρούς κανόνες για την εξυγίανση, περισσότεροι όροι για τις τράπεζες για να γίνεται ε, δυνατή η εξυγίανση. Αυτή η, ε, τώρα η όρεξη έχει μειωθεί και γι' αυτό το συζητήσαμε το θέμα και με ανταλλαγή επιστολών και με ερωτήσεις και αμφιβάλλομαι πολύ ότι τα σχέδια εξυγίανσης που διαπραγματευτήκατε με τις αντίστοιχες ε, ε, οντότητες ε, είναι σωστές και ένομες διότι δεν έχουν τους σωστούς στόχους ούτε προβλέπουν δεσμευτικά μέτρα για να ξεπεράσουν τα εμπόδια στην εξυγίανση. Είπατε μέχρι το 2020 θα ολοκληρώσετε τα πλήρη δεσμευτικά σχέδια εξυγένσης για όλους τους οργανισμούς. Καλό θα ήταν να επιλέξετε μια ταχύτερη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, σημαντικό είναι για μας να μην πυροβολείτε τον αγγελιοφόρο. Ε, αυτό που κάνετε δεν αφορά τόσο πολύ τις δικές σας αρμοδιότητες και τη δική σας ετοιμότητα ανάληψης δράσης. Ε, θα ήθελα όμως ε, τώρα να εκφράσω την απογοήτευσή μας ε, που δεν υπάρχει ανάληψη μεγαλύτερης ε, δέσμευσης από εσά. Να προσπαθήσω να απαντήσω. Για τον Banco Popular και εγώ πολλές φορές ε, εκπλήσωμαι από ε, τις πάρα πολλές ε, πτυχές του προβλήματος. Ε, εντάξει, ε, είχαμε πολλές, ε, μια, μια χιονοστιβάδα προσφυγών, αγωγών που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Λογικό. Βεβαίως έγινε πολύ θόρυβος. Χρειάζεται. Ας το κρίνουν αυτοί που έκαναν το θόρυβο. Τώρα, για τη μείωση της όρεξης ενίσχυσης των κανόνων, εμείς όπως και παλιά θέλουμε να εφαρμόζουμε τους υφιστάμενους νόμους και να φροντίζουμε να μπορεί να λειτουργήσει η εξυγένση των τραπεζών. Ε, τα, τα, τα προγράμματα δεν τα διαπραγματευόμαστε με τις τράπεζες. Εμείς, είναι δικά μας σχέδια. Πρέπει όμως να ακούσουμε τις τράπεζες την άποψή τους και να βεβαιωθούμε ότι λαμβάνουν τη σωστή δράση και ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Πολύ θα ήθελα να αναλάβω δέσμευση για μια ταχύτερη διαδικασία. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να πω ότι όπως κάναμε και για τα MRL το 2017 αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο και ουσιαστικό βήμα για τις μεγάλες τράπεζες. Η δεύτερη κατηγορία ακολουθεί και να είστε βέβαιοι ότι θα ακολουθήσουμε την ίδια πορεία και με τα, για να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια και τα συνεφή. Για τα εμπόδια πάντοτε θα πρέπει να κάνουμε κάποιους ελιγμούς, γιατί δεν θέλουμε να σταματήσουμε το έργο της, εξυ... της δυνατότητας εξυγίανσης. Πρώτα θα πρέπει να λύσουμε το πρώτο ε, πρόβλημα, ίσως ε, και πολλές φορές να δουλέψουμε μέσα σε τρία επίπεδα παράλληλα. Να είστε βέβαιοι ότι την εντολή μας την παίρνουμε πολύ στα σοβαρά. Πολύ θα ήθελα να μπορώ να δηλώσω ότι το 2019 θα ολοκληρώσουμε, αλλά δεν θέλω να ε, υποσχεθώ υπερβολικά πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Catch η ΕΝΕΦ, η FTD δεν βλέπω. Ο κύριος Φερνάντες έχει το λόγο. Καλό σας απόγευμα, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ. Θα ήμουν ευτυχής να σας υποβάλω ερωτήσεις για το πρόγραμμα εργασίας του 18 και το πολιετές ε, πλαίσιο εργασίας, αλλά δεν παραμένει χρόνος. Γι' αυτό θα σας μιλήσω για την περίπτωση του Banco Popular. Τέσσερις ερωτήσεις. Είπατε ότι οι πληροφορίες από το Reuters διέρευσαν και κατά κάποιο τρόπο ε, διεύρυναν τις δηλώσεις σας στο Bloomberg, διότι ε, στην περίπτωση του Bloomberg εσείς δεν αναφερθήκατε ρητά στην Banco Popular, αλλά στην απάντησή σας αναγνωρίσατε ότι συμπεριλαμβάνεται στην ανάλυση σας την Banco Popular. δηλαδή ότι θα έπρεπε να γίνει ε, μία εξυγίανση. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να γίνει σχόλιο ούτε για τη ΜΕΝ ούτε για τις δε τράπεζες. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιες διαρροές στο μέλλον ή σε μελλοντικές συνεντεύξεις πώς μπορούμε να αποφύγουμε ε, κάτι τέτοιες ε, ατυχείς ε, δηλώσεις. Για την Deloitte, στις δύο εκθέσεις, ελέγχθη ότι δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν για λόγους ασφάλειας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι μετά την εξυγίανση υπήρξε μεγάλη αστάθεια στην αγορά εξαιτίας ακριβώς αυτής της ε, χρηματοοικονομικής αστάθειας. Γι' αυτό θεωρώ ότι τουλάχιστον οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να μπορέσουν να μελετήσουν αυτές τις εκθέσεις και σε μελλοντικές περιπτώσεις τέτοιες εκθέσεις περί εξυγίανσης θα έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Ως προς την κατάρτιση αυτής της ε, εξπόστ έκθεσης ε, της ε, Deloitte. Εσείς ε, μιλήσατε για την αποφυγή συγκεκριμένων συγκρούσεων συμφερόντων, αλλά εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Δεν κατανοούμε γιατί αυτός που καταρτίζει την πρώτη έκθεση καταρτίζει και τη δεύτερη. Εδώ υπάρχει πραγματικά σύγκρουση συμφέροντος. Θα ήθελα στο μέλλον να λάβετε υπόψη ότι αυτή η σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες ως προς τη σταθερότητα των αγορών και της κατάστασης των ε, τραπεζών. Η τέταρτη ερώτηση αφορά την Τραπεζική Ένωση. Εσείς είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, μία υποστήριξη έτσι ώστε να μπορέσει να δράσει το ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης στην Τραπεζική Ένωση. Θα αρχίσω με την πρώτη ερώτηση σε σχέση με την ε, διαρροή πληροφοριών από το Bloomberg. Μπορείτε να κάνετε ό,τι διασυνδέσεις θέλετε, αλλά ε, ρωτήθηκα από ένα δημοσιογράφο για το ε, θέμα της Banco Popular και τη μείωση της αξίας της μετοχής της, αλλά εγώ είπα ότι η Banco Popular είναι, συγκαταλέγεται σε μια κατηγορία τραπεζών που μας απασχολούν. Δηλαδή αυτό επακριβώς ανέφερα. Δεν οδήγησα σε περαιτέρω συζητήσει για την Banco Popular. Για την έκθεση Deloitte ε, διαφωνώ ότι υπήρχε αστάθεια στις αγορές μετά την εξυγίανση στη Banco Popular που έγινε αποδεκτή και από τους ε, Ισπανούς συναδέλφους. Δηλαδή ότι δεν υπήρξε καμία επίπτωση ως προς το κύριο χρέος ή τις τράπεζες. Πολλοί είπαν τι συμβαίνει, αναρωτήθηκαν τι συμβαίνει με αυτή την τράπεζα, αλλά δεν υπήρξε θέμα ε, χρηματοοικονομικής ε, σταθερότητας. Ως προς την έκθεση Deloitte, είπαμε πολλές φορές ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστές αξιολογήσεις και θέλουμε να ε, γίνεται η εκτίμηση από τον ίδιο φορέα. Ε, δεν μπορώ να αποκλείσω ότι αυτό θα γίνει και στο μέλλον ή εάν ανακύψουν λόγοι θα υπάρχουν δύο ξεχωριστοί ε, αξιολογητές. Για μένα φαίνεται λογικό να γίνεται κάτι τέτοιο. Αν λάβουμε υπόψη την πληθώρα ε, αξιολογητών. Όπως, όσο αφορά την διαφάνεια, θα προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο να δημοσιοποιήσουμε τα στοιχεία αξιολόγησης της Deloitte που δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και θα ενταχθούν, θα αναρτηθούν στον ιστό τοπό μας, αλλά θα αφορά μόνο το, ε, ε, το θέμα της, ε, των στοιχείων που δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Ως προς το EDs και την εξυγίαση θεωρώ ότι υπάρχει και ε, το θέμα της εγγύησης δανειοδοτήσεων μέσα στα πλαίσια της εξασφάλισης και των καταθέσεων και θα δούμε τι θα γίνει μετά την αμοιβεοποίηση. Τώρα, το κατά πόσο το ίδις ε, θα, ε, αποτελεί, θα έχει μια άμεση συνδεσιμότητα, αυτό θα το, θα το αποφασίσετε εσείς ως νομοθέτης. Νομίζω ότι η Επιτροπή θα προτείνει το backstop και για την και για την ε, και στην περίπτωση του ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης. Καλώς ήρθατε. Έχω δύο σύντομα ερωτήματα για εσάς, λίγο στρεμόσα. Και σας εύχομαι βέβαια και κάθε επιτυχία στην, ε, σε επόμενες χρονιές ε, στο έργο σας. Πολύ Σύντομα λοιπόν στα αγγλικά. Το πρώτο ερώτημα, τι μπορούμε να μάθουμε από την υπόθεση Banco Popular, ίσως την επόμενη φορά που μια τράπεζα σταλεί ε, στο ενιαίο Συμβούλιο έξυγεσης, μπορεί να μην χρειαστείτε 48 λεπτά για να αποφασίσετε, αλλά 48 ώρες που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες ε, ή τέλος πάντων να υπάρχουν κανόνες για τις κυβερνήσεις κτλ αν αυτό σας βρίσκει σύμφωνο, τι έχετε να πείτε και για την έκθεση Deloitte. Αν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζητήσει την πλήρη έκθεση Deloitte, το Συμβούλιο σας θα τη δώσει. Ευχαριστώ. Απάντηση είναι πολύ απλό. Το Συμβούλιο Εξεγίανσης φυσικά και ακολουθεί ε, τις βουλές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αν δηλαδή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταλήξει αυτό το συμπέρασμα, θα ζητήσω για μια ακόμη φορά από τους δικηγόρους μας ε, να μου πούν την άποψή του, αλλά σίγουρα εμεί θα πρέπει να εφαρμόσουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Επίση και σε ό,τι αφορά τι ε, ποινέ και τα τα μελετάμε και στην προκειμένη. Και για την έφεση. Ε, θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Είναι ένα ε, θέμα λεπτό. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ζήτημα για τα 48 λεπτά. Όχι, δεν ήταν 48 λεπτά, όλη τη νύχτα μας πήρε. Δεν ήταν 48 ώρες βέβαια. Και ένα από τα επιχειρήματα ήταν πως σε περίπτωση που μια τράπεζα μέσα στη μέση της εβδομάδας καταρρεύσει, καλό θα είναι να έχουμε σε έσχατη λύση το μορατόριου ε, για τις αρχές εξυγίανσης. Αυτή είναι μια πρόταση επιτόπου, ε, επιτάπητο, συγγνώμη, υπάρχουν πολλά υπέρ και κατά που θα πρέπει να λάβουν υπόψη, όμως είναι ένα εργαλείο αυτό θα μπορούσε να μας βοηθήσει να φτάσουμε από μια τρίτη, μια τετάρτη στο Σαββατοκύριακο, έτσι να κερδίσουμε χρόνο, αν απαντώ στο ερώτημά σας. So, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. και για την πολύ καλή διοργανική συνεργασία που έχουμε. Συμβούλιο Εξήγησης και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω και το επόμενο αυτό βήμα να βελτιώσει την συνεργασία μας, να υπάρξει στον ατόμο περισσότερη διαφάνεια σε αυτά τα στοιχεία. Δεν αποκλείεται από ό,τι κατάλαβα στο μέλλον το δεχόμενο να έχουμε διαφορετικές εκθέσεις <coughs> με διαφορετικές οντότητες, διαφορετικές φορείς να δημοσιοποιούν εκθέσεις για να έχουμε και τη συνέχεια του διαλόγου θα δούμε, θα ψηφίσουμε βέβαια στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την παρουσία σας στην ακρόαση αυτή. Θα κάνουμε τώρα ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για να προσέλθουν οι βουλευτές και θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία και θα ψηφίσουμε βέβαια και για την ε, εκλογή της κυρίας Κένικ.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

Chair, can we vote? Λοιπόν, να ψηφίσουμε κύριε Πρόεδρε. Αλλά να κάνουμε και μια δοκιμή. Άρχεται η ψηφοφορία, δοκιμαστικά. Λείπουν 29, 30, 33, ελάτε. Ελάτε εδώ με τις κάρτες σας. Ε, αγαπητοί βουλευτές, ελάτε και καθίστε. Still, I, I still see... Ακόμα λείπουν. Okay. Okay, so the test is closed. Πέρας του της δοκιμής. Ωραία. Πάμε. Πρώτη ψηφοφορία. Είναι ο διορισμός της Elke König επαναδιορισμός δηλαδή ως πρόεδρος σε μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με τον κανονισμό όπως με όλους τους διορισμούς. Συν πράσινο ναι, κόκκινο όχι, άρχεται η ψηφοφορία, η αποχή είναι αποχή. Vote Πέρας. 31 υπέρ 9 κατά 0 αποχές. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε, επέτυχε ο επαναδιορισμός, συγχαρητήρια. Προχωρούμε. Σχέδιο οδηγίας για την ηλεκτρονική κάρτα θα έχουμε ονομαστική ψηφοφορία για την πρώτη τροπολογία. Γιατί αν εγκριθεί θα απορριφθεί η πρόταση, άρχεται η ψηφοφορία. Ζήτησε κάποιος το λόγο. Όχι. Ε, αυτή είναι η οδηγία. Η οδηγία. Είμαστε στην οδηγία. Πρώτα θα πιάσουμε την οδηγία. Και άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Άρα η πρόταση απορρίπτεται και καταπίπτουν τα πάντα. Τώρα θα κάνουμε το ίδιο και για τον κανονισμό. Ίδια διαδικασία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας το ίδιο. 24 υπέρ, 16 κατά χωρίς αποχές. Απορρίπτεται και ο κανονισμός. Η πρόταση καταπίπτει. Σχέδιο έκθεσης για πρόταση οδηγία για την προληπτική αναδιάρθρωση κλπ. κλπ. 117 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 118 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 119. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Συγγνώμη γιατί δεν φαίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 120 υπέρ. Κατά. Και πάλι έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται γιατί ισοψήφισαν. 121 και 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 123 υπέρ κατά έλεγχος συγγνώμη άρχεται η ψηφοφορία ψηφίζουμε την 123 Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 124 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά περίεργη πολιτική συσχετισμή έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. την 125. Άλλοι δύο να ψηφίσουν πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική α υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 18. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 129. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 130. Υπέρ Κατά. Έλεγχο στην 130. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Λοιπόν, 130 ήταν αυτή. Πάμε στην 131 υπέρ. Κατά μου φαίνεται η ίδια πλειοψηφία, αλλά θα ελέγξουμε την 131 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Α, δεν ήταν το ίδιο. 132 υπέρ. Κατά. Η πράσινη κατά. Απερίφθη λοιπόν. Ε, τροπολογία 20 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 133 υπέρ κατά η η υπέρ άρχεται η ψηφοφορία πολλαπλή συνδυασμή εδώ πέρας αλλά απερίφθη λοιπόν αυτή ήταν τώρα πάμε στην 21 Τώρα, υπέρ της 21, κατά αποχές δεκτή, 134 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 135. Και οι δυο κατά, ΕΛΚ και σοσιαλιστές. Όχι, γιατί σηκώσατε το χέρι σας εσείς και δείξατε καταψήφιση. Ο Μπράιν ψήφισε με την περβάνωση. Ε, η καρδιά σας είναι αριστερά. Άρχεται η ψηφοφορία. Βλέπω εγώ το χέρι σας να ακολουθεί. Λοιπόν, ε, ε εγκρίνεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Ε, δεν, όχι σαφώς εγκρίθηκε, αλλά εγκρίθηκε τέλος πάντων. 135 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία πέρας απερίφθη 137 υπέρ κατά αποχές έλεγχος μου φαίνεται ότι απερίφθη αλλά να βεβαιωθούμε Να ψηφίσουν και άλλοι δύο. Πέρας. Όντως απερίφθη. Με μικρή διαφορά. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 139 υπέρ. Ε, όχι, όχι. Όχι, όχι, δεν την ψηφίσουμε γιατί είναι ταυτόσιμη. 140 υπέρ. Κατά. Μου φαίνεται ότι απερίφθη, αλλά θα ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρασε. Απερίφθη. 22. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Στην 22 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 23. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ψηφίσουμε την 23 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 142. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική B υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία Θέλετε να κάνουμε ηλεκτρονική. Α, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Δύο ακόμη να ψηφίσουν. Πέρας. Πέρας. Δεκτή. Οπότε πάμε στην 151. Υπέρ. Κατά. Τους πράσινους δεν βλέπω. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 151. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, δώσε τον προσανατολισμό εκεί με τα χέρια. Δύσκολη, δύσκολο να δω πώς συμπεριφέρεστε. Πέρασε. Απερίφθη. 152 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 153 υπέρ. Κατά έλεγχος. Ψηφίζουμε την 153. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η ισοψηφία κατά ε, ε, περίφθη 172 υπέρ. Έλεγχος 172. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ξανά ισοψηφία, ξανά περίφθη. 156 υπέρ. Κατά έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 28. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Μου φαίνεται ότι εγκρίνεται, αλλά να βεβαιωθούμε. 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Περβάνς, είπες όχι, αλλά ψηφίζει υπέρ. Πέρας. Ξεκάθαρα εγκρίνεται. Γι' αυτό υπήρχε σύγχυση προηγουμένως. 154 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ψηφίζουμε την 154. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ξανά ισοψηφία απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ψηφίζουμε την 155. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 158 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ κατά νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά θα ελέγξουμε την 157 άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή 159 υπέρ Κατά. Έλεγχος. ψηφίσουμε την 159. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Πάλι η ισοψηφία απερίφθη. Συμβαστική C. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 169 υπέρ. Κατά Έλεγχος. με 169. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Με διαφορά μιας ψήφου. 168. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψηφίζουμε 168. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Πάλι ψηφία πάλι απορρίπτεται. Συμβαστική D, υπέρ. Με προφορική τροπολογία από τον εισηγητή, μάλιστα. Ψηφίζουμε προφορική τροπολογία. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Νομίζω. Αλλά θα το ελέγξουμε. Δεν ήταν απόλυτα σαφές. Ψηφίζουμε την 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. 173 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 174. 174-176 υπέρ. Κατά έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ισοψηφία. Πάλι. Απορρίπτεται. 178 υπέρ. Κατά. Τι κάνουν οι σοσιαλιστές, είναι υπέρ ή κατά. Υπέρ, μάλιστα. Και το ΕΛΚ υπέρ. Την 178, ε, δεκτή. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν βλέπω του CCR. Άρχεται η ψηφοφορία. Δείξτε το προσανατολισμό. Πέρας απορρίπτεται 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές έλεγχος νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά θα το ελέγξουμε ψηφίζουμε την 33 λοιπόν πέρας Απερίφθη με διαφορά μιας ψήφου. 188 υπέρ, κατά, οι σοσιαλιστές υπέρ, σωστά, αποχές εγκρίνεται, 189 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 190 υπέρ κατά έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 191 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική ή υπέρ κατά αποχές δεκτή. 199 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 200 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 202 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 203 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 204 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία πέρας Απορρίπτεται. 205 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 206 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 207 υπέρ κατά έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία τη 207. Πέρας απορρίπτεται με διαφορά μιας ψήφου 208 υπέρ κατά αποχές δεκτή 209 υπέρ κατά έλεγχος στη 209 άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή 212 υπέρ κατά αποχές δεκτή 213 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.14 υπέρ κατά έλεγχο στη 214 ψηφίζουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας απερίφθη με μια ψήφο διαφορά 215 υπέρ κατά αποχές ΕΛΚ 215 τι λέτε υπέρ μάλιστα δεκτή 216 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. 216 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 217 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. 217 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 218 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 219 υπέρ. Κατά. η πιλελεύθεροι είστε υπέρ της 219, 219. Δεκτή. 220 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 221 υπέρ. Κατά έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική F υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 228 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 229 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 230 υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 231 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 232 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να βεβαιωθούμε. Πέρας. Δεκτή με μια ψήφο διαφορά. 233 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 234 υπέρ κατά έλεγχος 234 ψηφίζουμε τη 234 πέρας απερίφθη 235 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος 235. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απερίφθη. 236 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 237 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 36 υπέρ κατά έλεγχος ε, την 36 δώστε για τους, προ... κατευθύνσεις των ομάδων <clears throat> πέρας δεκτή 238 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά έλεγχος 37 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Δεκτή. 239 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. 239. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απερίφθη. 240 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. 240. Άρχεται η ψηφοφορία. υπέρας. Απορρίπτεται. 241 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 242 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 243 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 244 υπέρ. Κατά κατά αποχές απορρίπτεται 245 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 246 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 247 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 248 υπέρ κατά αποχές δεκτή 249 υπέρ κατά Έλεγχος στη 249 έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 250 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 252 υπέρ. Κατά. Α, καταπίπτει 251. Έλεγχος 252. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη 252. Πέρας. Δεκτή. 253 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. 253 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Έλεγχος 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική G υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 258 υπέρ. Κατά Έλέγχο 258 μου φαίνεται ότι απορρίπτεται αλλά δεν βλέπω καλά τα χέρια πέρας απορρίπτεται ε, με μικρή διαφορά 259 υπέρ κατά έλεγχος 259 άρχεται η ψηφοφορία πέρας Ισοψηφία απορρίπτεται. 260 υπέρ. Α, όχι, έχει αποσυρθεί. 261. 261 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Ήταν υπέρ τη σοσιαλιστές 261, μάλιστα. 262 υπέρ, κατά έλεγχος στη 262 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας δεκτή. 263 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 264 υπέρ κατά έλεγχος. 264 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 265 υπέρ κατά έλεγχος. 265 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 266 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. 266. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με μια ψήφο διαφορά. 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή 267 υπέρ κατά αποχές έλεγχος μου φαίνεται απορριπτικά αλλά έλεγχος παρόλα αυτά ψηφίζουμε 267 πέρας απερίφθη 268 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 269 υπέρ. Κατά έλεγχος. 269. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, μάλιστα, εσείς είσαστε υπέρ. Μάλιστα. Συγγνώμη, δεν σας είδα. Πέρας. Δεκτή. 270 υπέρ. Κατά. Έλεγχος 270. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 45 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβιβαστική H υπέρ κατά αποχές δεκτή Δεκτή 274 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική ΑΙ, υπέρ κατά αποχές δεκτή. 282 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 283 υπέρ κατά έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας δεκτή. Ε, J με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή 292 υπέρ κατά έλεγχο στη 292 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 56 και 70 όχι και 60 υπέρ Κατά. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτές. 293. Όχι. Καταπίπτει. Καταπίπτει. 57 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 58 υπέρ κατά έλεγχο στην 58. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 59 υπέρ κατά. Ε, ελέγχουμε. Την 59. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 2,96 υπέρ Κατά. Έλεγχο στη 296. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ισοψηφία απορρίπτεται. 295 υπέρ. Κατά. Έλεγχο στη 295. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 297 υπέρ κατά έλεγχος 297 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 298 υπέρ κατά αποχές δεκτή 200, ε, όχι, συμβαστική και υπέρ κατά αποχές δεκτή, τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβαστική L υπέρ κατά αποχές δεκτή, τροπολογία 67 υπέρ κατά έλεγχος, 67, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, απορρίπτεται, 68 υπέρ, 68 υπέρ, κατά, Έλέγχο Είναι 68. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 69. Υπέρ. Κατά αποχές. Απο... Ε, ε, ναι. Η συμβαστική M υπέρ κατά αποχές δεκτή. 1 ε, ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Την τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 74 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 75 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική ο υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 78 υπέρ κατά έλεγχο, στην 78 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας δεκτή. Συμβαστική πι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 83 υπέρ κατά έλεγχος 82-83 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτονται τροπολογία 7 υπέρ κατά τι λέει το ΕΛΚ κατά είναι του 7 απορρίπτεται 84 υπέρ κατά Έλέγχο στην 84 άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή Εμείς ψηφίσαμε την 84, εσείς να πάτε τώρα να ελέγξετε την 7. 7. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία την 7. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική Q υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 88 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. 88 άρχεται η ψηφοφορία. πέρας δεκτή 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική R υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές έλεγχος στη 10 έρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Δεκτή. Η 96 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 98 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ κατά αποχές έλεγχος στην 100 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές δεκτή 102 υπέρ κατά έλεγχος στην 102 άρχεται η ψηφοφορία πέρας. Απορρίπτεται 103 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Α, νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα το ελέγξουμε. Δεν είδα τους πράσινους. Πέρας. 104. Πέρας. Απερίφθη με μια ψήφο διαφορά 105 υπέρ κατά αποχές δεκτή 106 υπέρ κατά έλεγχος στην 106 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται συμβαστική S υπέρ κατά αποχές δεκτή Προπολογία 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική Τι υπέρ κατά αποχές δεκτή, τροπολογία 14 υπέρ κατά η φιλελεύθερη υπέρ έλεγχος. Όχι, όχι, όχι έλεγχος. Εγκρίνεται. Αν είστε υπέρ, εντάξει. 112 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά Έλεγχο στη 15 άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή η 114 υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 115 υπέρ υπέρ κατά αποχές δεκτή 116 υπέρ κατά έλεγχος ψηφίζουμε την 116 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται με μια ψηφοδιάφορα διαφορά ψηφίζομαι ονομαστική ψηφοφορία την πρόταση όπως τροποποιήθηκε άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. 33 ε, υπέρ 2 κατά 4 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ωραία. Τέλος. Το κείμενο το τελευταίο. Όλο μαζί. Πρέπει να ψηφίσουμε όλο μαζί. Όλο. Όλο. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Τροποποιη... τροποποιημένο ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Δεκτό, 33 υπέρ, μια ψήφος κατά και τρεις αποχές. Ευχαριστώ. To pass the chair now. Τώρα θα δώσω το, την Προεδρία, θα την αναλάβει κάποιος άλλος.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 Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, τελικά δεν έφυγα. Δεν είναι η μέρα αυτή η συνηθισμένη, αλλάζουν ε, συνεχώς τα πράγματα και τα δεδομένα. Ε, Έχουμε περίεργες πολύπλοκες εξέλιξεις. Λοιπόν, θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ σήμερα τον κύριο Μάσιμο Μπορντινιόν, που είναι μέλος του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Δημοσιομικού Συμβουλίου, ήρθε δεχόμενος ε, την πρόσκλησή μας για να συμμετάσχει στη σημερινή ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη τη Επιτροπή ΕΚΟΝ εκπροσωπεί τον καθηγητή Τάγκεσεν, ο οποίος δυστυχώς δεν μπόρεσε να αποτεχθεί την πρόσκλησή μας λόγω μιας ε, αλλαγής της τελευταίας στιγμής ε, στη μέση διάταξη του Eurogroup και εκεί μιλά αυτή τη στιγμή για το ίδιο θέμα που θα μας απασχολήσει εμά. Είχαμε βέβαια ήδη μια ανταλλαγή απόψε με τον καθηγητή Τάγκησεν τον Ιούλιο μετά τον διορισμό του, οπότε και είχε έρθει σε μια συνεδρίαση τη Επιτροπή ΕΚΟΝ και μα ενημέρωσε για τι απόψει που έχει το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για σημαντικά σημεία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Στι 15 Νοεμβρίου το Συμβούλιο δημοσίευσε την πρώτη της έκθεση και εκεί αναφέρεται ο τρόπος εφαρμογής ε, του δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τονίζονται οι ατέλειες και αναφέρονται τα περιθώρια βελτίωσης. Θα ακούσουμε τον κύριο Μπονιόν να μας κάνει μία εισαγωγική παρέμβαση και εν συνεχεία θα ακολουθήσει ο γύρος ερωταπαντήσεων τους ευρωβουλευτές. Κύριε Μπονιόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του Νίλ Στάγκεσεν αλλά και του Συμβουλίου Γέννη Θέλω να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης, ε, την οποία, όπως είπατε και εσείς, ε, δημοσιοποιήσαμε στις 15 Νοεμβρίου. Και ελπίζω όλοι να έχετε λάβει αντίγραφο αυτής της έκθεσης. Αλλιώς μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας. Τι λέει αυτή η έκθεση λοιπόν. Ορίστε, εδώ τα βλέπετε, ελπίζω τουλάχιστον, μπορείτε να τα δείτε. Τι κάνει τη σχέση έκθεση ουσιαστικά. Παρουσιάζει ε, μια ανάλυση της εντολής ε, του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Τι είναι το πρώτο πρέπει να κάνουμε είναι να αξιολογήσουμε την εφαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης. Και αυτό γίνεται στο τμήμα 2. Εστιάζουμε στο τμήμα 2 στο 2016, αυτή τη χρονιά, είναι το τελευταίο έτος που μπορούσαμε να δούμε ένα πλήρη κύκλο εποπτείας σε ό,τι αφορά ε, τη συμβουλές που μας έδωσαν ε, για το φθινόπωρο από το τον Οκτώβριο μέχρι και την Άνοιξη του 2016. Πρέπει να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι νέος ε, οργανισμός. Ουσιαστικά τέλη του 2016 συσταθήκαμε, άρα φέτος, του Μαρτίου, φέτος το Μάρτιο ξεκινήσαμε τις εργασίες μας. Στην ουσία αυτή είναι η πρώτη μας αιτήσια έκθεση και θα παρουσιάζουμε συναλέγραφα και κάθε χρόνο αυτή την αιτήσια έκθεση. Το δεύτερο που ε, περιλαμβάνει η εντολή μας ως βασικό καθήκον είναι η συνεργασία μας με τα εθνικά δημοσιονομικά συμβούλια ιδίω για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Και αυτό κάνω στο τμήμα 3 του με αναφορεωμένο στην ανάλυση των ανεξάρτητων δημοσιονομικών φορέων μετά το δημοσιονομικό σύμφωνο του 2012. Κάποιες χώρες είχαν τέτοιους θεσμούς, κάποιες δεν είχαν. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση εστιάζουμε σε δύο πολύ σημαντικές ε, και ενοφανεί ε, τέτοιους φορείς, τον Ιρλανδικό φορέα, και τον Δανέζικο, που όμως έχει πιο μακρόχρονη ιστορία από πίσω. Επόμενο καθήκον μας είναι παροχή συμβουλών στην Κομισιόν για τον καλύτερο δυνατό δημοσιονομικό προσανατολισμό για την Ευρωζώνη. Και αναδρομικά και προοπτικά. Δηλαδή, αναδρομικά σε σχέση με το τι έγινε το 2016, στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή, οι συμβουλές της Κομισιόν προς τα κράτη-μέλη. Τι... Πώς εφαρμόστηκαν από τις χώρες και συνολικά από την Ευρωζώνη αλλά και προοπτικές συμβουλές παρέχουμε για το δημοσιονομικό προσανατολισμό για το 2018. Αυτό ήδη έγινε τον Ιούνιο του 2017 σε ένα ξεχωριστό έγγραφο. Τέλος παρέχουμε προτάσεις ε, για τη μελλοντική εξέλιξη του δημοσιονομικού πλαισίου στο τμήμα 5 της έκθεσης συγκεκριμένα. Αυτή λοιπόν είναι η δομή, αυτή είναι η διάρθρωση της έκθεσης. Έτσι είναι οργανωμένη. Ποια είναι τα βασικά μηνύματα. Το πρώτο μήνυμα είναι ότι αν δει κανείς προς τα πίσω και σε ό,τι αφορά το 2016 αλλά και τα τελευταία χρόνια θα διαπιστώσει ότι ήταν δύσκολη χρονιά, δύσκολες χρονιές για αυτούς που χαράσουν τις δημοσιονομικές πολιτικές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο γιατί υπήρξαν στιγμές, ιδίως μετά τη μεγάλη κρίση που ναι υπήρξε ανάκαμψη σε κάποιες χώρες Άλλε φορές πιο ε, μεγάλη, άλλες φορέ πολύ λιγότερη. Υπήρχε χαμηλός απληθωρισμός ε, και υπήρχε και το ιστορικό της κάθε χώρας και θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και συγκεκριμένα τι έπρεπε να γίνει βλέποντας τη μακροοικονομική κατάσταση να χαλαρώσουμε τους κανόνες τους δημοσιονομικούς δηλαδή αυτό όμω θα μπορούσε να υπονομεύσει τη βιωσιμότητα μακροπρόθεσμα των δημόσιων ή να ακολουθήσουμε την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή να εφαρμόσουμε αυστηρά του κανόνε. Αυτό βέβαια έχει το πρόβλημα που θα μπορούσε να υπονομεύσει την ανάκτηση που εξακολουθούσε να είναι εύθραυστη, ιδίω το 2016. Και το γενικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε και εφαρμόσαμε με διακριτική ευχέρεια και ευελιξία το Σύμφωνο Σταθέτης και Ανάπτυξης με αποτέλεσμα να θετήσουμε έναν δημοσιονομικό προσανατολισμό σε επίπεδο ευρωζώνη που θεωρούμε ότι ήταν το ενδεδειγμένο, αλλά όχι σε εθνικό επίπεδο. Υπήρχαν χώρε οι οποίε χρειάζονταν μεγαλύτερη σταθεροποίηση, άλλε βιωσιμότητα και αντιστρόφως. Ενώ άλλε χώρε αντίθετα, χρειάζονταν περισσότερη βιωσιμότητα και όχι σταθεροποίηση. Ένα άλλο συμπέρασμα είναι ότι οι κανόνες ε, είναι πολύπλοκοι. Γιατί υπήρξαν αρκετές αλλαγές. Και η διακριτική ευχέρεια βέβαια έπαιξε ρόλο. Ήταν πολύ ε, σημαντική η διακριτική ευχέρεια και η κρίση το γεγονό ότι δεν ναι χρειάζεται διεκδικηθεί για την εφαρμογή των κανόνων, αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένη συγκεκριμένε διατάξει. Το θέμα είναι να μπορεί να υπάρχει διαφάνεια και προβλεψιμότητα για να αντισταθμίζεται η κατάσταση λόγω του πολύπλοκου των κανονισμών. Να υπάρχει δηλαδή διαφάνεια. Ένα γενικό λοιπόν συμπέρασμα του τμήματος 2, το οποίο επαναλαμβάνουμε και στο τμήμα 5, είναι ότι αν θέλουμε να κοιτάξουμε προς το μέλλον υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης και εντός του τρέχοντος πλαισίου, δηλαδή μπορεί να γίνει κάτι ήδη στο τρέχον πλαίσιο χωρίς να χρειαστεί να γίνουν μεγάλες αλλαγές στο νομοθεσία στη συνθήκη, αλλά και εκτός αυτού, πέραν αυτού. Πώς τα πήγαμε τώρα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερής και Ανάπτυξης του 2016. Αν δείτε τι λέει η Κομισιόν, τα δημοσιονομικά σχέδια δηλαδή που υπευλήθησαν το 2015 η Κομισιόν ε, εκεί μίλησε ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν προβλήματα μη συμμόρφωσης με διάφορες χώρες. Και για το προληπτικό σκέλος και για το διορθωτικό σκέλος. Πάντως τελικά είδαμε ότι υπήρξε συμμόρφωση μπορεί να υπήρχε κίνδυνος, ε, το 2015 έτσι αντιλαμβανόμασταν τα πράγματα, αλλά το 2017 η κατάληξη της Κομισιόν είναι ότι τελικά υπήρξε συμμόρφωση. Και αυτό δεν οφείλεται τόσο πολύ στη μεγάλη οικονομική μεγέθυνση. Γιατί αυτή λίγο πολύ ακολούθησε τις εκτιμήσεις που είχε κάνει η Κομισιόν το 2015 ήταν μάλιστα χαμηλότερη ονομαστική ανάπτυξη για τα πολύ χαμηλότερα τα επίπεδα του πληθωρισμού από τα αναμενόμενα. Όμως ο κύριος της μη συμμόρφωσης αντιμετωπίστηκε ιδίω με τη διακριτική ευχαίρεια και τη μεγαλύτερη ευελιξία. Και επίσης κάποιες χώρες που δεν συμμορφούντο μιλάω για το διορθωτικό σκέλος εδώ, πήραν περισσότερο χρόνο και ακυρώθηκαν οι ποινές τους, οι κυρώσεις τους. Μιλώ ιδίω για την Ισπανία και την Πορτογαλία. Άρα, η γενική κατάληξη, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι ναι, μην υπήρξαν ατέλειες, θα σας δώσω περισσότερες ε, εξηγήσεις προς αυτό, ατέλειες λοιπόν ε, του συμφώνου, αλλά δεν υπήρξαν σοβαρά σφάλματα. Και καταλήγουμε εμείς στο ε, συμπέρασμα ότι είναι καλύτερο να έχουμε κανόνες που εφαρμόζονται έστω και ατελώς από το να μην εφαρμόζονται ή από το να έχουμε μια μεγάλη χαλάρωση ή πολύ αυστηρή εφαρμογή. Νομίζουμε λοιπόν ότι ήταν η καλύτερη εξέλιξη αυτή. Ποιες είναι οι περιπτώσεις ατελούς εφαρμογής. Τα βλέπετε βέβαια πιο αναλυτικά στην έκθεση. Δεν θα, τα, δεν θα μακρηγορήσω. Για το προληπτικό σκέλος, για παράδειγμα. Δύο δείκτες πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την νομοθεσία για να αξιολογηθεί αν υπάρχει κίνδυνος απόκληση. Η διαρθρωτική ισορροπία και οι δαπάνες. Θεωρητικά θα έπρεπε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά επειδή μετρώνται διαφορετικά, δεν συμπίπτουν πάντα. Οι επιπτώσεις μπορεί να έχουν. Άρα θα πρέπει κανείς να κρίνει και να αποφασίσει Ποιο είναι ο σωστός δείκτη να χρησιμοποιήσει. Και είδαμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις η επιλογή για το κατα... γιατί προτιμήθηκε ο ένα δείκτη από τον άλλο δεν ήταν ε, συνεπής ανά χώρα ή συν χρόνο. Είχαμε επίση άλλα θέματα. Οι ρήτρε ευέλιξε για την Ιταλία, τη χώρα μου. Η πληξιμότητα βασίζεται ουσιαστικά στην υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά αυτό εξολογείται εκ των υστέρων. Δεν ήταν σαφές όμως τελικά αν υπήρξε απόφαση της Κομισιόν για το κατά πόσον έγιναν ή δεν έγιναν οι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. στα τα συνταξιοδοτικά. Επίσης έχουμε διαδικασίε προβολικού ελλείμματο για Ισπανία, Πορτογαλία. Εδώ υπήρξε κάποια καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την αφορμή τη διαδικασία ε, το Μάιο του 2016 είχε πει ότι δεν προχωρούν ε, σωστά τα πράγματα η Κομισιόν, αλλά μετά από δύο-τρει μήνε ζήτησε παράταση των προθεσμιών και αυτό δεν συμφωνούσε με ορισμένε στάσει του Συμβουλίου. Επίση, σε κάποιε χώρε δεν είχαμε επαρκή μείωση του χρέου. Δεν κινήθηκε όμως κάποια διαδικασία. Λόγω της χρήσης αυτών των άλλων συναφών παραγόντων πέραν του κανόνα του χρέους και η ονομαστική ανάπτυξη το 2016 σε κάποιες από αυτές τις χώρες ήταν πολύ μικρή. Και αυτό βέβαια δημιουργεί πρόβλημα. Δεν μπορεί να μειωθεί το ονομαστικό χρέος εύκολα. Και βέβαια είχαμε και άλλα προβλήματα με τις υπηρεσιακέ κυβερνήσεις. Τι γίνεται όταν έχεις μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Τι μπορεί να και τι μπορεί να κάνει μια τέτοια κυβέρνηση. Αυτό το συζητήσαμε. Τώρα, ποια είναι η κατάσταση με το δημοσιονομικό προσανατολισμό έκανε κάποια καθοδήγηση, πρόσφερε κάποια καθοδήγηση το 2015 η Κομισιόν το Συμβούλιο. Ουσιαστικά να είναι ουδέτερη ω ομοδοποιημένο αυτό ο προσανατολισμό και να υπάρχει διαφοροποίηση σε εθνικό επίπεδο. Για του λόγου που ανέφερα προηγουμένω και θα βρείτε πολύ περισσότερη τεκμήρωση στην έκθεση. Εύθραυστη ανάκαμψη, υπήρχε ο κίνδυνο ύφεση και σε χώρε. Κάποιες χώρες ήταν πολύ ψηλά τα επίπεδα χρέους. Αυτό ήταν πρόβλημα και η νομισματική πολιτική είναι περιοριστική. Είχαμε φτάσει στον πάτο. Δεν μπορούσαμε να πέσουμε κάτω από το μηδέν στα επιτόκια. Τι γίνεται λοιπόν με αυτή τη μακροοικονομική κατάσταση. Ένα ότερν έγινε, όπως λέμε. Ακολουθήθηκε ένας επεκτατικός δημοσιονομικός προσανατολισμός Είχαμε θετικό ισοζύγιο δρατικό. Δεν ήταν όμως βέλτιστη κατάσταση αναχώρα. Σε κάποιες χώρες ο κίνδυνος βιωσιμότητας ε, ήταν ε, μεγαλύτερος και δεν εφάρμοσαν όλες τις απαιτήσεις. Βέβαια θα μπορούσε να είναι πιο στριπτική η πολιτική αυτή αν υπήρχε χώρος Ε, Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το Σύμφωνο σταθερότητα και Ανάπτυξης θα πρέπει να οδηγήσει σε μία ε, ισόμετρη ανάπτυξη. Αλλά σε χώρες που υπάρχει η υπερβολική απόδοση θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούν να υπάρχουν υψηλότερες δαπάνες. Και η ΟΝΕ ναι βασίζεται σε μία κοινή νομισματική πολιτική αλλά εθνική φορολογική πολιτική. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ορισμένες ε, περιπτώσεις, να το δούμε το ζήτημα κατά περίπτωση, αλλά δυστυχώς ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να δούμε την ανεξάρτητη, τις ανεξάρτητες δημοσιονομικές αρχές της χώρες. παρατηρούμε ότι αυτή η ανεξάρτητη αρχή λειτουργεί καλύτερα σε χώρες που έχουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής. Και σημασία έχει και η συμμόρφωση με αυτές τις ε, δημοσιονομικές αρχές και φυσικά έχει σημασία να δούμε κατά πόσο υπάρχει διαφορά μεταξύ της αποτίμησης της κυβέρνησης και της ανεξάρτητης ε, δημοσιονομικής αρχής και στο τέλος η κυβέρνηση θα πρέπει να συμμορφωθεί αν δεν συμμορφωθεί να επεξηγήσει γιατί. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μεταρρύθμιση των εθνικών αρχών και οι κυβερνήσεις να επέμβουν εγκαίρως. Με βάση τα σχόλια των ανεξάρτητων δημοσιονομικών αρχών, ποιες προτάσεις κάνουμε σε σχέση με το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας ορισμένες προτάσεις είναι απλές και δεν σημαίνουν μία μεγάλη αλλαγή στην ε, νομική βάση. Αυτό που κάνουμε και προτείνουμε είναι να άρουμε τις ασυμμετρίες που υπάρχουν. Δηλαδή, στα πλαίσια του συμφώνου υπάρχει ασυμμετρία μεταξύ των καλών και κακών καιρών και του διορθωτικού σκέλους σε σχέση με το προληπτικό σκέλος. Προσπαθούμε λοιπόν να μειώσουμε αυτές τις ασυμμετρίες και ο στόχος είναι μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης, της ανάκαμψης, μία χώρα να αφήσει ικανό χώρο για δράση ως προς την βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. Και επίσης οι κυρώσεις δεν είναι αποτελεσματικές. Δηλαδή οι επικρίσεις που ακούτε σε σχέση με το σύμφωνο ε, σταθερότητας και ανάπτυξης είναι ότι δεν είναι αποτελεσματικό. Δεν συμφωνούμε γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει ένας κυρωτικός μηχανισμός. Όμως, από την άλλη πλευρά, είναι δύσκολο να επιβάλλει κανείς κυρώσεις σε ένα κράτος που είναι κυρίαρχο. Άρα θα πρέπει να αντικαταστήσουμε τις κυρώσεις με κάποιο είδος ερεσιμότητας, δηλαδή όταν δεν τηρούνται ορισμένες ευρωπαϊκές ε, δαπάνες, ιδιαίτερα ως προς τα διαρθρωτικά ταμεία, γιατί τα διαρθρωτικά ταμεία δεν είναι σημαντικά για όλες τις χώρες, τότε θα πρέπει να ε, αυξήσουμε την ερεσιμότητα και εάν επιθυμούμε περισσότερη ε, δημοσιονομική ε, δυνατότητα, ικανότητα, τότε θα πρέπει και πάλι να υπάρχει αιρεσιμότητα. Πολύ περισσότερο από τις κυρώσεις. Επίσης, προτείνουμε να συνδέσουμε αυτά τα δύο τμήματα, δηλαδή το σύμφωνο και την διαδικασία μακροοικονομικής εξισορρόπησης. Προτείνουμε λοιπόν να ορίσουμε τους μέσο και μακροπρόθεσμους στόχους με βάση τις μακροοικονομικές ανισότητες. Και υπάρχει και το θέμα του πολυσχηδούς χαρακτήρα του εγχειρήματος και της διαφάνειας, γιατί εδώ ε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αλλαγή των συνθήκων, αλλά να απλουστεύσουμε τους κανόνες που είναι ιδιαίτερα περίπλοκοι και υπάρχουν και πολλοί κανόνες και ε, έκτακτες ανάγκες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη με βάση συγκεκριμένες ε, ε, ρήτρες διαφυγής. Αυτές οι ρήτρες διαφυγής ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο όταν υπάρχει παροχή συμβουλών από κάποια ανεξάρτητη αρχή. Και στη συνέχεια η Επιτροπή και το Συμβούλιο αποφαίνεται. Επίσης μιλάμε για την ε, λειτουργία της σταθερότητας στα πλαίσια της ΟΝΕ. Ε, δεν έχετε πολύ χρόνο, λέει ο Πρόεδρος. Προσπαθήστε να ε, ολοκληρώσετε. Με συγχωρείτε, δεν έλεγξα το ρολόι μου. Εδώ λέμε λοιπόν ότι υπάρχουν προβλήματα στο, στην ΟΝΕ, γι' αυτό θα πρέπει ε, να είμαστε πιο ανθεκτικοί μέσα στα πλαίσια των συμμετριών ημί και φυσικά ε, αυτό που έχει σημασία είναι να εστιάσουμε την προσοχή μας στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι περισσότερες προτάσεις δεν έχουν οριστεί επακριβώς Μιλάμε για έναν ε, ε, μηχανισμό προστασίας και παράλληλα ένα σχέδιο, ένα επενδυτικό σχέδιο. Και θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται ένα σχέδιο προστασίας των επενδύσεων. Κάτι το οποίο είναι μια πιο πιστική εναλλακτική γιατί ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη και στην ζήτηση. Θα σταματήσω εδώ. Ήδη σας είπα τι συνέβη, αλλά τα αποτελέσματα είναι τα ίδια με αυτά που σας προανέφερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση και για την έκθεση σε σχέση με το Ευρωπαϊκό ε, Δημοσιονομικό Συμβούλιο Πρόκειται για κάτι το απόλυτα σαφές, αλλά υπάρχει, υπάρχουν πολλές ε, περιπλοκότητες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και υπάρχουν ε, και πολλές ατέλειες. Υπάρχει ένας υψηλός βαθμός ατελειών του συστήματός μας και γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε τη σωστή η εξισορρόπηση μεταξύ προβλεψιμότητας και ενός θεσμικού πλαισίου το οποίο θα πρέπει να ορίσουμε γιατί έχουμε να κάνουμε με κυρίαρχα κράτη με κοινούς κανόνες οι οποίοι κανόνες όμως έχουν ένα ειδικό στάτους και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε πώς η Επιτροπή θα φτάσει σε μία εξισορρόπηση τα τελευταία χρόνια. Ε, κάτι το οποίο ε, δεν είναι τέλειο, αλλά εν πάση είναι λιγότερο ατελές από άλλα πλαίσια που είχαν προβλεφθεί. Ακόμα και η ατέλεια μπορεί να αποτελεί μία σοφή εξορρόπηση, όπως ορίζουν τα πέντε παραδείγματα που μας ε, δώσατε και γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Εμείς ως Κοινοβούλιο είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε σχέση και με τα προνόμια που διαθέτουμε και το θέμα ενέχει πολλές περιπλοκότητες και από πλευράς συμμετοχής των Εθνικών Κοινοβουλίων. αλλά φυσικά ο ρόλος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου είναι ε, ύψης της σημασίας. Ο συνάδελφος από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Έκπληξη. Το ΕΛΚ δεν είναι εδώ. Εγώ συμφωνώ με τον Πρόεδρο που λέει ότι είναι ισορροπημένη η έκθεση Ευχαριστούμε και για την παρουσίαση και για την έκθεση. Θυμήθηκα ότι η Κομισιόν είχε σύσταση. Αυτή είναι η πρώτη ερώτησή μου δηλαδή. Σύσταση για Γερμανία και Ολλανδία. Και με επενδύσεις 50 δις. Και αυτό συμφωνεί με το δικό σας συμπέρασμα. Ότι η δημοσιονομική θέση ήταν καλή, αλλά όχι σε επίπεδο κάθε χώρας. Πρέπει να ε, έκανε μια πρόταση η Κομισιόν που την ευθυγραμμίζεται, αλλά πώς μπορούμε να κάνουμε πιο συμμετρικούς τους κανόνες Έχουμε μια, ένα παράδειγμα, μια καλή πρόταση της Κομισιόν που όμως αγνοήθηκε από τα κράτη-μέλη. Και το ευρύτερο ερώτημα, γιατί λέτε για απλούστευση κανόνων, ταχύτητα επίτευξης μεσοπρόθεσμων στόχων. Ποια είναι η ισορροπία. Μιλάτε για επιβολή απλούστευση κανόνων, αλλά και για δημοσιονομική ικανότητα σε κεντρικό επίπεδο. Και λέτε ότι θα υπήρχε μεγαλύτερη σταθερότητα αν υπήρχε ένα κεντρικό δημοσιονομικό όργανο. Όμως, όταν χτυπήσει η επόμενη κρίση ή η ύφεση, πάλι θα είμαστε αβοήθητοι έτσι όπως είμαστε τώρα. Πολλές χώρες δεν μπορούν σε αποκεντρωμένο επίπεδο να κάνουν επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Οπότε συνολικά τι είναι το πιο σημαντικό, η αποκεντρωμένη, η κεντρική η δημοσιονομική οντότητα ή η απλούστευση και η εφαρμογή των κανόνων τι μετράει πιο πολύ στη ζυγαριά. Ελπίζω ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να μας δίνει εναλλακτικέ και επιλογές, αλλά να θέτει και βασικά ερωτήματα κέρια για τη σταθερότητα της Ευρωζώνης. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω ακόμα, δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά επειδή έχω εργαστεί στην Ολλανδία σε κεντρικό επίπεδο σχεδιασμού για περίπου 10 χρόνια αναρωτιόμουν τι διδάγματα αντλήσαμε. Δεν ξέρω, διαβάζοντας την έκθεση. Εγώ από την τράπεζα είδα ότι ο αντίκτυπος πολλαπλασιάζεται όταν δίνουμε εναλλακτικές στους πολιτικούς. Ε, ε όχι, εναλλακτικές δίνουμε, δεν δίνουμε συμβουλές. αυτό είναι το σωστό. Ε, δεν θεωρούμε ότι η τράπεζα θα είναι διαμφισβήτητη στην άποψή τη, ε, όχι βέβαια, αλλά θα... Ε, πολλές τράπεζες έχουν καλή φήμη με την έννοια ότι δίνουν εναλλακτικέ. Αυτές τις δύο ερωτήσεις είχα να σας κάνω. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. μπορώ να ομαδοποιήσω κάποιες ε, ερωτήσεις. Χρειαζόμαστε πιο απλούς κανόνες και πιο κεντρική δημοσιονομική ικανότητα. Για να αρχίσω με την πρώτη ερώτηση, ναι, έχουμε ένα πρόβλημα στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξη όπως είναι τώρα, γιατί μια χώρα η οποία ξεπερνά τους μεσοπρόθεσμους στόχους δεν, έχει τη νομική δεν, δεν τελεί υπό νομική υποχρέωση. Δεν υπάρχουν εργαλεία δηλαδή για να την πιέσετε να δαπανά περισσότερο. Η πρόταση που λέει ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα συντονισμό των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών, αλλά και δεν έχουμε μεγάλο αποτέλεσμα. Στην περίπτωση που αναφέρατε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει, ναι, έκανε πρόταση στην Γερμανία και την Ολλανδία να, δαπανούν, να αυξήσουν τις δαπάνες. Αλλά δεν αποκολουθήθηκε η πρόταση από τις δύο χώρες. Υπάρχει ασυμμετρία. Πώς θα λυθεί η ασυμμετρία? Μια πιθανή λύση, ένας τρόπος δηλαδή να πάμε να βρούμε λύση, είναι με κάποια ικανότητα δημοσιονομική κεντρική. Αν μια χώρα δηλαδή αποφασίσει ότι για πολιτικούς λόγους και προτιμήσεις δεν θέλω να αυξήσω τις δαπάνες μου, ε, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνουν και πολλά ενάντια σε μια τέτοια απόφαση. Αν έχετε όμως μια κεντρική δημοσιονομική ικανότητα, ένα νέο φορέα, εκεί μπορεί να βοηθηθεί το πρόβλημα και να λυθεί. Στην Ευρώπη, στη συζήτηση που γίνεται τώρα, δεν μιλάμε, μιλάμε για τον ευρω, ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ενωσιακό, αλλά δεν μιλάμε για μεγάλο, σαν ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Κάνουμε κάποιες προτάσεις να υπάρχει ένας στηρικτικός, σταθεροποιητικός μηχανισμός σε περίπτωση ασύμετρων ε, σοκ, αλλά ε, αυτό θα είναι καλύτερο από το τίποτα σε ό,τι αφορά την στήριξη. Γι' αυτό στηρίζομαι αυτές τις, ε, ε, αυτά τα προγράμματα προστασίας των επενδύσεων. Γιατί σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στις χώρες που επλήγησαν πιο πολύ από την κρίση, ο τρόπος ε, που αντέδρασαν οι ε, ε, είναι να μειώσουν τις επενδυτικέ δαπάνε. Αυτό είναι πιο εύκολο σε πολιτικό επίπεδο, αλλά αυτό θα βλάψει, θα κάνει μεγάλη ζημιά μέσω αλλά και βραχυπρόθεσμα, γιατί είναι μικρότερη ζήτηση και μακροπρόθεσμα μειώνεται η δυνατότητα ανάπτυξης. Αυτό λοιπόν ε, χρειάζεται πιο πολλές προσπάθειες. Ως Μάσιμο στο Συμβούλιο ε, επικεντρωνόμεθα σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μιλάμε για τη δημοσιονομική ικανότητα γιατί αυτό αφορά πιο πολύ την εντολή μας σε γενικότερο επίπεδο. Αν με ρωτάτε όμως τι χρειάζεται για να γίνει πιο ανθεκτική η Ευρωζώνη, η δημοσιονομική ικανότητα, η κεντρική, είναι ένα από τα πράγματα που χρειάζονται. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση, και η Κεφαλαϊκή Ένωση, η Ένωση Κεφαλαίων κλπ. Χρειάζονται περισσότεροι μηχανισμοί για να δώσουν κάποια διασφάλιση. Ε, αλλιώς ε, διατρέχουμε κίνδυνο, συμφωνώ μαζί σας, να ακολουθήσει ένα άλλο σοκ και να βρεθούμε εμείς χωρίς κανένα όπλο στα χέρια μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο, ο κύριε Στραμόζα. Μια σύντομη ερώτηση. Μετά από δέκα χρόνια ε, μετά την έναρξη της κρίσης είδαμε σε κάποιες χώρες δημόσιο χρέος πάνω από 3%, πάνω από το όριο 3% και βλέπουμε τώρα τους επόμενους μήνες ότι η νομισματική πολιτική θα ξαναγυρίσει στην ομαλότητα και δεν θα, ε, θα υπάρξει αύξηση των επιτοκίων και οι δημοσιονομικές δαπάνες θα αυξηθούν στις χώρες αυτές. Οι μηχανισμοί κυρώσεων βλέπουμε ότι δεν ε, έχουν αποτέλεσμα. Πώς θα γίνουν λοιπόν οι δημοσιονομικοί κανόνες πιο αποτελεσματικοί σε ενωσιακό επίπεδο ή δεν υπάρχει καμιά ελπίση. Τι εννοείται με τον ε, ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Εννοείται τον... Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει ο δημοσιονομικός κανόνας και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός ο δημοσιονομικός κανόνας, αυτή είναι η δικιά μας η πρόταση. Ε, για την πρόβλεψή σας θα πω ναι, ελπίζω ότι εξομαλύνονται οι καταστάσεις και τώρα η οικονομική κατάσταση βελτιώνεται σε πολλές χώρες, οπότε ήρθε η ώρα να, να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε και να αναδιοργανώσουμε τις δομές για να λειτουργούν καλύτερα. Και πώς θα λειτουργήσουν καλύτερα. Καταρχήν πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τώρα ήρθε η ώρα για μια χώρα όπως η δική μου που έχει πολύ υψηλό χρέωση ή άλλες χώρες που έχουν μεγάλο έλλειμμα να προσπαθήσουν να μειώσουν τις δαπάνες διότι εκεί το κόστος θα είναι χαμηλότερο. Ε, οικονομικά θα λέγαμε ότι αυτή είναι η ώρα όπου θα πρέπει να δημιουργήσουμε ε, κάποιες, κάποιο, ε, κάποιες ζώνες ασφαλείας για το μέλλον. Ε, και προβλέπονται κάποιοι τέτοιοι μηχανισμοί. Χρειάζεται μια διακριτική ευχέρεια η οποία θα λαμβάνει υπόψη διαφορετικά πράγματα. Αν έχετε δηλαδή κύκλο θετικό ή αρνητικό στον προϋπολογισμό, δημοσιονομικό κύκλο. Αυτό πρέπει να το κάνουμε καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Μια δημοσιονομική πολιτική τι πρέπει να είναι, τι περιμένουμε. Θα ε, πρέπει να δίνει αρκετούς πόρους στήριξης της οικονομίας όταν πλήττεται από αρνητικά σοκ. Και αντίθετα, αντίστροφα. Ε, στην Ευρωζώνη οι περισσότερες ε, δημοσιονομικές πολιτικές είναι προκυκλικές και έκαναν περισσότερα λάθη με την έννοια ότι ε, δεν βελτίωσε τον κύκλο, τον έκανε, τον, τον, τον, έκανε, τον όξινε. Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή που πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα για τον έλεγχο των δαπανών και τη μείωση του χρέους. Ο δημοσιονομικός κανόνας τα επιτρέπει αυτά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μπορούμε να μειώσουμε τις ασυμμετρίες και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να λειτουργήσει ακόμα περισσότερο ο μηχανισμός που έχουμε. Ναι, είναι δύσκολο να αρχίσουμε να, να πούμε ότι τώρα μπήκαμε σε περίοδο καλή. Ακόμα υπάρχουν ε, φαινόμενα υστέρησης, ε, επενδυτικά κενά Υπάρχει δηλαδή έλλειμμα επενδύσεων και υπάρχουν διαφορετικές τάσεις και ε, ε, φυγόκεντρες δυνάμεις. Ε, σίγουρα όμως είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από ότι όταν είμαστε σε ύφεση υπερβάνους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Α, ξέχασα. Περβά, συγγνώμη, ο κύριος Βιέγκα. δεν ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος. Είναι ασυνήθιστο να μην πάρει σαν τι πολιτικέ ομάδε που ξέχασα τελικά κάποιον. Μιγγέλη, συγγνώμη, ήσουν εκεί και δεν σε είδα. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πω στα πορτογαλικά. Και θα είμαι και σύντομο. Για να μπορέσουν να λάβουν το λόγο και άλλοι συνάδελφοι. Έχω δύο πολύ απλά ερωτήματα. Είχα και πιο πολλά, αλλά τέλος πάντων ε, θα περιοριστώ σε δύο. Το πρώτο ερώτημα αφορά την προστασία των επενδύσεων. Θα ήθελα να μας πείτε κάτι παραπάνω. Και η αποφυγή ε, της πολυπλοκότητας είναι κάτι σημαντικό. Θέλουμε δημόσιες επενδύσεις και να προωθήσουμε το σχέδιο Juncker. Αλλά αυτό θα οδηγήσει σε πολύπλοκη νομοθεσία και είναι αντίθετο με αυτά που μας προτείνετε εσείς και συστήνετε εδώ σήμερα. Το δεύτερο, τι γίνεται με τη διαδικασία οικονομικών ανισορροπιών και το ΠΕΣΕ. Εγώ βλέπω μια σχέση, αλλά επισήμως δεν ξέρω. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κανόνες ώστε το σύστημα να γίνει τελικά όμως και πιο πολύπλοκο. Hey, thank you very much. Ε, Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τα ερωτήματά σας. όταν έγιναν αυτέ τι προτάσει δεν ήταν πολύ συγκεκριμένε. Ήμασταν σε κάπω αμήχανη θέση και εμεί στο Συμβούλιο Δημοσιονομικό. Κατατέθηκαν κάποιε ιδέε στο έγγραφο τη Κομισιόν για την ε, δημοσιονομική ικανότητα. Αλλά δεν συζητήθηκαν επαρκώ προτάσει αυτέ ώστε να μπορούμε να κρίνουμε τα πράγματα. Θέλει περισσότερη επεξεργασία αυτή η πρόταση. Υπάρχουν ανάγκες η πρώτη είναι ότι οι επενδύσεις μειώνονται σε όλες τις χώρες. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό, για να προστατεύσουμε τις επενδύσεις. Δηλαδή το σχέδιο Juncker έχει αποδώσει, προοριζόταν όμως κυρίως για ιδιωτικές και όχι για δημόσιες επενδύσεις. Άρα πρέπει να προστατεύσουμε και τις δημόσιες επενδύσεις. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν διαφορετικές υποδείξεις. κάποιο ταμείο ε, που σε περίοδο παχιών αγελάδων ε, η χώρα βάζει κάποια κεφάλαια για περίοδο συχνών αγελάδων κτλ. κτλ χαμηλό επιτόκιο, αρκεί η χώρα να κρατάει χαμηλά ε, τα επίπεδα των δαπάνων κτλ. Απλά δεν έχουμε ακόμα επεξεργαστεί τις λεπτομέρειες. Η Κομισιόν και το Συμβούλιο όμω εργάζονται πάνω σε αυτό το θέμα και μα ικανοποιεί αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών στην Ευρώπη, έχουμε αυτά τα δύο συστήματα. Το ένα λειτουργεί, δηλαδή η Κομισιόν μπορεί να συσχετίσει τη συμπεριφορά της χώρας με τη δημοσιονομική συμπεριφορά. Και έχουμε αυτή την διαδικασία μακροοικονομικών ε, ανισορροπιών που υπάρχει μένα αλλά δύσκολα κινητοποιείται. Πρέπει να κάνουμε τη σχέση μεταξύ μακροοικονομικής έκβασης και κυβερνητικής συμπεριφοράς. Άρα, εμείς νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διασυνδέσουμε αυτά τα δύο μεταξύ τους περισσότερο αν θέλουμε να εγγυηθούμε τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, δεν πρέπει τόσο να ελέγχουμε τις δημόσιες πάνε στο δημόσιο χρέος, αλλά να προσπαθούμε να είναι πιο ανθεκτική οικονομία. Με τις μακρονομικές ισορροπίες, δηλαδή, και την εξάλληψή τους θα μπορούσαμε να πετύχουμε τη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να πούμε είναι ότι θα πρέπει η ταχύτητα, ο ρυθμός να ρυθμιστεί καλύτερα για την επίτευξη των μέσων προθεσμών στόχων με την κατάσταση μακροοικονομικών ανισορροπιών. Μια χώρα που έχει παραδοσιακά ισορρεύσει πλεόνασμα μπορεί να θέλει να καθυστερήσει την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων, των μάλλον στόχων. Μπορεί να υπάρχουν και άλλε δυνατότητε. Εμεί θεωρήσαμε όμω ότι αυτή είναι μια καλή λύση. Ίσως να περιπλέκει πράγματα πράγματα. Δεν νομίζω όμως ότι θα είναι τόσο μεγάλο το βάρος. Είναι σχετικά εύκολο. Υπερβάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσίασή σας και για την συμμετοχή σας σε αυτή τη συζήτηση σε μια περίοδο που είναι επίκαιρα αυτά τα θέματα κατά κάποιο τρόπο. Ο ρόλος σας είναι να παρακολουθείτε την κατάσταση καθημερινώς, μια νέα δομή, είστε ένας νέος φορέας, ταυτόχρονα όμως όλα τα θέματα τα οποία σχολιάσατε είναι αντικείμενο προβληματισμού ακόμη μεταξύ των κρατών μελών αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα το πρώτο μου συγκεκριμένο ερώτημα είναι κατά πόσον είχατε κάποια συμμετοχή, δώσατε τη γνώμη σας σε αυτόν τον προβληματισμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς συνεργάζεστε με τις εθνικές αρχές. Αυτό το δίκτυο μεταξύ εθνικών αρχών πώς λειτουργεί για την ανταλλαγή πληροφοριών, διαγνώσεων και σκέψεων για το μέλλον. Μιλήσατε για την πολυπλοκότητα του Δημοσίου Συμφώνου, την είναι κατάλαβε κανείς τους στόχους κτλ. Αυτά τα συζητούμε εμείς στο Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων και εδώ και καιρό. Υπάρχει μια πρόταση. Δεν την αναφέρατε νομίζω. Και ουσιαστικά είναι η θέση του Κοινοβουλίου. Είναι ευρεία αποδοχή στο Κοινοβουλίο. Δηλαδή, αντί να έχουμε δυσνόητους κανόνες και να είναι δύσκολο να υπάρξει οικειοποίηση σε αυτό το επίπεδο, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα λεγόμενο κώδικα σύγκληση. δηλαδή στόχου σύγκληση προ τα πάνω. Θα ορίζονται σε ευρωπαϊκή κλίμακα, σε καθαρά παραδείγματος χάρη, τους μισθού, τις επενδύσεις, διοικητικές ικανότητες κτλ. Και θα υπάρχει και ένα οδικό χάρτη που θα καταρτίζεται σε εθνικό επίπεδο. Με πενταετή χρονικό ορίζοντα, για παράδειγμα. Αυτό το έχετε συζητήσει. Και τέλο πάντων, όπω και αν έχει, ποια είναι η άποψή σα από αυτού. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή στη συζήτηση έμεσα. Βεβαίω υπάρχει συνεχιζόμενη συζήτηση με την Κομισιόν, την Αρμόδια Γενική Διεύθυνση, για ανταλλαγές απόψεων και πληροφοριών αλλά δεν συμμετέχουμε άμεσα στις συζητήσεις. Εμείς ε, συζητήσαμε την πρόταση για την Ευρωζώνη και η αντίδρασή μας ποια είναι. Εμείς ε, ε, στηρίξαμε το επίσημο έγγραφο. Αν η Κομισιόν δηλαδή κάνει προτάσεις όπως αυτή την πρόταση που θα παρουσιαστεί στις 6 Δεκεμβρίου. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Αν η πρόταση αφορά την εντολή μας, την εντολή του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, οπωσδήποτε πρέπει να την εξετάσουμε. Αλλά δεν συμμετείχαμε άμεσα στις συζητήσεις. Για τις εθνικές δημοσιονομικές αρχές, ναι, έχουμε σχέση μαζί τους και πρέπει να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο αλλά υπάρχει μια διεθνής οργάνωση ε, τρόπων των δημοσιονομικών αρχών και τουλάχιστον ε, δύο φορές το χρόνο συναντώνται και στις δύο περιπτώσεις ε, εμείς πήγαμε να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας και να συζητήσουμε μαζί τους. Στην έκθεσή μας προτείνουμε ότι ο ρόλος των εθνικών αρχών στην εποπτεία ε, θα πρέπει να ε, στηρίζεται και να γίνεται περισσότερη συζήτηση με την Κομισιόν. Μια συγκεκριμένη πρόταση αφορά την υποστήριξη της πρότασης της Κομισιόν για ανεξάρτητη τεχνική ε, γνωμοδότηση. Τέλος, για τον ε, κωδικά σύγκλησης δεν θα απαντήσω. Θα μου επιτρέψετε. Πρέπει να ξέρουμε περισσότερα στοιχεία, περισσότερες λεπτομέρειες και μετά θα συζητήσω με ευχαρίστως. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που έχουμε εξετάσει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου ως θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε εδώ την ανταλλαγή απόψεων. Θέλω να ε, ευχαριστήσω τον κύριο Μπορδινιόν για την ε, παρουσία του και για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση και τον διάλογο ο οποίος θα συνεχίσει, βεβαίως θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμεθα με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο Τη Δετάρτη περιμένουμε μια πρόταση από την Κομισιόν η οποία ενδιαφέρει και το Κοινοβούλιο και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και ελπίζω ότι η συνεργασία μας θα συνεχιστεί και θα ε, βεβαίως θα εξετάσουμε εντελεχέστερα την έκθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης ε, σχέδιο γνωμοδότησης του συναδέλφου Ραμόν Τρεμόσα. Είναι ένα σχέδιο γνωμοδότησης για την Επιτροπή Μεταφορών που θα ψηφίσει το Μάρτιο την έκθεσή της. Κύριε Ισηγητά, έχετε τον λόγο για να μας παρουσιάσετε το σχέδιο γνωμοδότησης. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τη γνωμοδότησή μου σε σχέση με τη γνωμοδότηση του κύριου Μάρκου Πίπερ στην Τραν. Πρόκειται για ένα θέμα αερομεταφορών που σχετίζεται και με θέματα ανταγωνισμού. Γι' αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας. Εμείς ως Επιτροπή και πολλά μέλη σε τακτά ε, χρονικά διαστήματα θέτουμε αυτό το θέμα στην Επίτροπο Φερστάκεν. Μιλάμε για την αναθεώρηση του κανονισμού 868 και νομίζω ότι θα πρέπει να βελτιωθεί. Θεωρώ ότι το έγγραφο της Επιτροπής είναι πάρα πολύ καλή βάση συζήτησης. Ξέρετε ότι έχω αντιταχθεί στις κρατικές επιδοτήσεις τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει αναδιάρθρωση έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός στον τομέα των παγκοσμίων αερομεταφορών. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει δημοσιονομική ε, διαφάνεια όταν πρόκειται για επιδότηση ιδιαίτερα των τρίτων χωρών. Θεωρώ ότι ο ανταγωνισμός θα πρέπει να είναι ίσος και δίκαιος. Θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη με το Συμβούλιο και ιδιαίτερα ορισμένα κράτη-μέλη που θέλουν να αποδυναμώσουν αυτή την πρόταση, καθώς και τις εξουσίες έρευνας της Επιτροπής. Νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει την διενέργεια ερευνών ως προς διακρίσεις που υπάρχουν από ορισμένες αερογραμμές. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ίσως παγκόσμιος ανταγωνισμός και δίκαιες πρακτικές, έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι κρατικές επιδοτήσεις όσο αφορά τους ευρωπαϊκούς αερομεταφορείς. Γι' αυτό και οι τροπολογίες μου μιλούν για δημοσιονομική Διαφάνεια. Επίσης, οι αερομεταφορείς θα μπορέσουν να παρέμβουν ε, εάν υπάρχει αμφισβήτηση. Επίσης, η περίοδος έρευνας θα πρέπει να μειωθεί από δύο σε ένα χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ για το ΕΛΚ. Θα δώσω το λόγο στο ΕΛΚ. Ε, θα ήθελα να πω ότι αναλαμβάνω την Προεδρία για διάφορους λόγους, αρχαιότητα κλπ. Ο Αλέν Λαμασούρ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αν αυτό ήταν το κριτήριο της αρχαιότητας, εγώ θα κατήχα τη θέση. Θα ήθελα εντάχει, όπως και ο εισηγητής, να πω ότι το ΕΛΚ συμμερίζεται την άποψή του και προσωπικά λυπάμαι που το 2004 που ήμουν στο Κοινοβούλιο, όπως και εσείς, κυρία Πρόεδρε, εγκρίναμε ένα κείμενο καθόλου ικανοποιητικό και Είχαμε πολλά δυσίωνα ε, ε, συμβάντα ε, ανάμεσα στους κοινοτικούς αερομεταφορείς και τους αερομεταφορείς τρίτων χωρών για να φτάσουμε σε ένα κείμενο το οποίο βελτιώνει σχετικά αλλά όχι ικανοποιητικά το προηγούμενο διατακτικό. Μπορούμε λοιπόν να υποστηρίξουμε τις τροπολογίες του εισηγητή και προτείνω με τους άλλους σκιώδεις να έρθουμε σε επαφή μαζί του για να δούμε κατά πόσο θα μπορούσαμε να έχουμε ε, περισσότερο ευρω... ένα περισσότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργίας για τους σοσιαλιστές. Ο κύριος Συμπαγέ θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να χαιρετήσω την πρόταση της Επιτροπής που θέλει να υποστηρίξει τους ε, ε, Ευρωπαίους αερομεταφορείς από πολιτικές διάκρισης από τρίτες ε, χώρες. Μιλάμε για 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 500 δις στο κοινοτικό ΑΕΠ. Γι' αυτό θα πρέπει να, να προστατεύσουμε τους ευρωπαϊκούς αερομεταφορείς έναντι τρίτων χωρών για να έχουμε ίσους όρους ανταγωνισμού. Βεβαίως δεν πρέπει να είμαστε και αφελείς, διότι θα πρέπει να, υπάρχει, ε, να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθίσταται σαφές ότι δεν θα πρέπει να δεχόμαστε ε, τις κρατικές επιδοτήσεις ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ούτε και εκτός αυτής. Σε σχέση με τον κανονισμό του 2004 που δεν εφαρμόστηκε ποτέ, η Επιτροπή προβάλλει αλλαγές για αυτό το modus operandi ως προς την αντιμετώπιση των πολιτικών διάκρισης, ενώ ο οργανισμός του 2004 μιλούσε για ε, οικονομικές ε, πολιτικές, φορολογικές πολιτικές που οδηγούν σε διάκριση. Μιλούσαμε ήδη από το 2004 για τη δυνατότητα προσφυγής των αερομεταφορέων. Χρειάζεται λοιπόν αναθεώρηση του κειμένου και θα προτείνω και εγώ ορισμένα στοιχεία γιατί η Ευρώπη θα πρέπει να προστατεύει περισσότερο τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενούς της όταν αντιμετωπίζουν αυτές τις μορφές διάκρισης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν βλέπω άλλους σκιώδεις να είναι παρόντες εκτός και αν κάποιος κρύβεται, φαίνεται πως όχι. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελαν το λόγο. Φαίνεται πως όχι. Ξέρω ότι η Γενική Διεύθυνση MOVE εκπροσωπείται από τον κύριο Ντουσάρ. Δεν ξέρω κατά πόσο θέλει να παρέμβει. Ναι, απλώς για να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησής του καθώς και την επιθυμία του να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα του κειμένου. Και θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας προς την ίδια κατεύθυνση με εσάς για αυτό το πολύ σημαντικό ε, κείμενο για τον ανταγωνισμό στην Ευρώπη και τη συνδεσιμότητα των περιφερειών. Ευχαριστώ πολύ. Εφόσον δεν ε, ζητά κανείς άλλο το λόγο, θα δώσω το λόγο στον εισηγητή που έχει όσο χρόνο θέλει για να σχολιάσει τα λεγόμενα των συναδέλφων. Ωραία, ωραία, πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ ε, τους για την υποστήριξή τους. Νομίζω ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε μια ευρεία πλειοψηφία και σε επίπεδο Συμβουλίου ως προς την υποστήριξη των αερομεταφορέων όλου του κόσμου και για τον τρόπο λειτουργίας ε, των αερομεταφορέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από αυτή την ε, συζήτηση, την εμπεριστατωμένη συζήτηση, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι στις 12 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Θα ε, εξετάσουμε τις τροπολογίες 24 Ιανουαρίου και θα ψηφίσουμε στις 21 Φεβρουαρίου του επομένου έτους, έτσι ώστε όταν αποφανθεί η Επιτροπή Μεταφορών στις 5 Μαρτίου να μπορέσει να λάβει υπόψη τη δική μας συνεισφορά. Τελειώσαμε με την Επιτροπή μας. Θα ήθελα όμως οι συνάδελφοι να παραμείνουν στην αίθουσα ή να επανέλθουν στις 18.30 γιατί τότε θα έχουμε μια κοινή συνεδρίαση με την ΛΥΜΠΕ κατά τη διάρκεια της οποίας θα εξετάσουμε με την Επίτροπο τον κατάλογο Eurova, δηλαδή των χωρών που δεν συνεργάζονται. Θα τα πούμε λίγο αργότερα.